Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες και σύντομα, διότι στις 10 έχουμε τον Επίτροπο που θα περιμένει στις... Και μετά πρέπει να... Έτσι πρέπει να τελειώσουμε τις ψηφοφορίες πολύ γρήγορα. The ε, ε, κύριε Μαγκίνες, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα την κατανόησή σας γιατί δεν έχω μαζί μου την κάρτα ψηφοφορίας μου οπότε μπορώ να σας να χρησιμοποιώ το χέρι μου για να ψηφίσω ε, πρόεδρος. Ναι, Μάρετ, μπορείτε να ζητήσετε από το προσωπικό σας, από τους υπαλλήλους σας να φέρω την κάρτα διότι ε, αργότερα θα έχουμε μια ψηφοφορία που θα διαρκέσει αρκετή ώρα. Ξεχνάμε με το σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης. Αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλου του 1998 για τους έμονους οργανικούς ρήπους. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Τροποποίηση του πρωτοκόλλου του 1998 για την διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρήπανση σε μεγάλη απόσταση από βαρέα μέταλλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Now we are Περνάμε στο σημείο 23 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση περί βελτίωσης τη καινοτομία και τη οικονομική ανάπτυξη στη διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του μέλλοντος. Ε, η ο κ. Τζόφολη. Να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία τη τροπολογία. 1 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρινέται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ας ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Όχι. Ζητά συγγνώμη ο πρόεδρος. Ε, περνάμε στη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 39 για την παραγραφό 4 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Avete votato tutti? Ψηφίσατε άπαντε. 39. Πέρα ψηφοφορία, Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Avete votato tutti. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Adottato. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 53 τμήμα 2 ως νέο κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Avete votato tutti? Ψηφίσατε άπαντες. Ακόμα όχι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ψηφίσατε άπαντες πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70 πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 70 τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Ψήφισατε πέρα στι ψηφοφορίε εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται 74 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές ε, να ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78, τμήμα 2, υπέρ. Κατά. Αποχές, έγκρινεται. Τροπολογία 83, υπέρ. Κατά. Αποχές, έγκρινεται. 84 υπέρ κανείς κατά ωραία είναι σαφές απορρίπτεται τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογία 98. με ε, ονομαστική ψηφοφορία ζητήθηκε από το EFDD 19 άτομα υποστηρίζουν το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Ποιος υποστηρίζει την ονομαστική ψηφοφορία, το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία δεν είστε 19, συγγνώμη. Ωραία, θα ψηφίσουμε να τεσχυρώ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία να περάσουμε τώρα στην τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 104 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Πέρας ψηφοφορία συγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή τον κύριο Τζόφολη. Περνάμε τώρα στην έκθεση Dennis Macker για την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα. Και ας ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία στην τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας, Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ανά το Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Τροπολογία 59. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε. Ψήφισατε άπαντες πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, είπα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αν θέλετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, να το ελέγξουμε για την τροπολογία 96. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε απαντέ, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 141 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. και η συνάδελφος Μαγκίνες ψήφισε με το καρτελάκι οπότε απορρίπτεται τροπολογία 135 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ψηφίσατε άπαντες πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 309, συγγνώμη, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 332, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 157, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 158, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 12 να το ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 161 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 165, υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε. Ξεφίσατε άπαντες πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες πέρα φοφορίας. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 176 υπέρ. Ε, συγγνώμη ο πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε την 176 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ψηφίσατε άπαντες πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται Να ψηφίσουμε τώρα την 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 220 υπέρ Συγγνώμη, 200. Τροπολογία 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 213. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 215. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 240 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. το Ψηφίσατε άπαντε, πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 229. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. βοτά το Ψηφίσατε άπαντε πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 250 τμήμα 2 υπέρ Ζητά συγγνώμη ο Πρόεδρος. Πρέπει να πάμε στην 259. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. «265 πρώτο τμήμα υπέρ» «Κατά» «Αποχές» «Εγκρίνεται» Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 271 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 278 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 280 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 276 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 2.77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Avete votato tutti, il voto... Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 285 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την 285. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 287 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 306 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 308 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 322 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 320 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. το Ψήφισατε άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 323 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποσύρεται. Όχι, μιλάμε για την 323, λέει ο πρόεδρος. Δεν αποσύρεται. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Τώρα. 324. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 327. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 320, 325. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 329 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογία 330 δεν ψηφίζεται 328 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 331 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 326 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε Avete votato tutti. Ψηφίσατε άπαντες. τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 336. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 338. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 345 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 346 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 21 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 353 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 350 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 352 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 354 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 362 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Avete votato tutti, il voto è chiuso. άπαντες, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογία 364, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 363, υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Avete votato tutti, il voto όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 366 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. 366 πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά θα το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της 365 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 367 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 368 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 369 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη Εγκρίθηκε. Τροπολογία 370. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 371. Υπέρ. Α, μια στιγμή. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε την 371. Καλύπτεται. Ψηφίζουμε την 372. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 373. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα σε τελευταίες σκέψεις. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω να σε ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Στη συνέχεια πάμε στην τροπολογία 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 19 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλώς. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Να ελέγξουμε. Καλώς, θα ελέγξουμε. Τροπολογία 20. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Α, πέρα τη ψηφοφορία. Ναι, βλέπω τα πράσινα φωτάκια στα έδρανά σα, γι' αυτό λέω ότι εγκρίθηκε. Σαφέ το αποτέλεσμα. Τα χέρια δεν φαίνονται καλά όταν τα σηκώνετε. Τροπολογία 22 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 36. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Όχι. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 4. Από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 4. Γιατί ο συμβασμός 16 δεν εγκρίθηκε. Υπέρ. Εγκρίθηκε, επειδή εγκρίθηκε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 32-32 το αποτέλεσμα. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Πρέπει να την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ΔΕΒΕ 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. ΔΕΒΕ 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίσουμε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις Εγκρίθηκε και συγχαρητήρια στον κύριο Ντεσμάκερ, στον εισηγητή. Πέτερλε. Ο κύριος Πέτερλε τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Πέτερλε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το νέο σύστημα καταλόγων ψηφοφορία. Ε, τα πράγματα έτσι είναι πολύ πιο σαφή και πολύ πιο γρήγορα. Και καλέ γιορτέ. Ευχαριστεί ο Πρόεδρο. Δεν έχει τελειώσει η συνεδρίαση. Στι 11 θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και στι 11 έχουμε τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Μιγγέλα Κανιέτε. as you wish. Dear colleagues, we have been... Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε εδώ με τον Επίτροπο, τον Μιγέλ Αρίας Κανιέτε και τον ευχαριστούμε που ήρθε, που βρισκόμαστε τόσο κοντά στα Χριστούγεννα, αλλά πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να ανταλλάξουμε απόψεις μετά τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στο Παρίτσι όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Χαιρόμαστε πολύ λοιπόν που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα του COP21 με τον Επίτροπο. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία νομίζω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι πολύ για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε στο Παρίσι, αλλά επίσης και επειδή έχουμε την ευκαιρία με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναμειχθούμε και εμείς μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Παρίσι. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία πρέπει να σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Επίτροπο για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα του δώσω όμως ευθύ αμέσως το λόγο για να κάνει την παρουσίασή του και μετά δίχως άλλο πολλοί συνάδελφοι θα ζητήσουν το λόγο για ερωτήσεις και για να συζητήσουμε παρετέρω κάποια θέματα. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ για να συζητήσω μαζί σα τα αποτελέσματα του COP21. Θέλω όμω να ξεκινήσω ευχαριστώντα την αντιπροσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχε στο COP21 υπό τον πρόεδρο ε, Τζοβάνι Λαβί και τον αντιπρόεδρο Ματίας Γκρότερ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ σας και για την ανεκτήμητη στήριξή σας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στο Παρίσι. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πάντα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κλιματική μας πολιτική. Ήσασταν ένα βασικό παίκτη για τι συζητήσει που γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά επιπλέον το έργο σα ήταν θεμελιώδη για τη διαμόρφωση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι που κάνει την πραγματική διαφορά για μια οικονομία χωρί άνθρακα και προκειμένου να παγιώσουμε την ηγετική μας θέση όσον αφορά την κλιματική πολιτική. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω όλους την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεργάστηκαν προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η συμφωνία αυτή. Την προηγούμενη εβδομάδα με ρωτήσαν κατά πόσο είμαι ευχαριστημένος ή όχι από τα αποτελέσματα που πετύχαμε στο Παρίσι και απάντησα ότι είμαι και χαρούμενος και ανακουφισμένος. Πρώτα απ' όλα γιατί τώρα έχουμε μια νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία η οποία θα μας δώσει τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από τους δύο βαθμούς. Είναι σαφώς ένα πολύ καλό μήνυμα προς τους επενδυτέ, τι επιχειρήσει, τους πολιτικούς και είναι μια στροφή η οποία έγινε και θα μείνει. Μετά από... και είναι ανεπίστρεπτη. Δεύτερον, γιατί μετά από πολλά χρόνια όπου η διεθνής κοινότητα δίσταζε για διάφορα γεωπολιτικά ζητήματα, στο Παρίσι καταφέραμε να ενώσουμε όλες τις χώρες του κόσμου υπέρ ενό κοινού σκοπού. Η συμφωνία είναι μεγάλο κέρδο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και δείχνει ότι η πολυμερή διάσταση εξακολουθεί να λειτουργεί όταν το διακύδευμα είναι παγκόσμιο, είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Και είναι και ένα σημαντικό μάθημα που πήραμε για τα επόμενα χρόνια και έτσι δώσαμε και νέα στα στην Έθνη. Και τρίτον, επειδή μετά από μια ταραχώδη χρονιά στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε μέλη κατάφεραν να δώσουν αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μείνωσε με μία, με μία ενωτική φωνή και μιλώντας έτσι με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε το άνισμα μέσω του οποίου οικοδομήθηκε μια ευρύτερη συμμαχία ή ύπατη συμμαχία φιλοδοξίας όπως τη λέμε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, στο Παρίσι αποκορυφώθηκε μια διαδικασία ετών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια οικονομική και πολυμερή συμφωνία για το κλίμα. Όταν ήρθα στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας πριν από τη διάσκεψη, κατέστησα σαφές ότι ένα επιτυχές αποτέλεσμα πρέπει πρώτον να είναι, έχει ένα μακροπρόθεσμο στόχο, δεύτερον να πρόκειται για μια περιοδική αναθεώρηση με ευελιξία ώστε να βάζουμε όλο και πιο φιλόδοξους στόχους κάθε φορά και τρίτον να ενισχυθούν οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας. Ε, η συμφωνία αυτή πέτυχε και τα τρία αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Για πρώτη φορά λοιπόν επιβεβαιώσαμε τον μακροπρόθεσμο στόχο διατήρηση τη μέση αύξηση τη θερμοκρασία παγκοσμίω κάτω από 2 βαθμού σε σύγκριση με την προβιομηχανική ε, περίοδο. Η Επιτροπή επίση καλωσορίζει την αναγνώριση που περιλαμβάνεται στη συμφωνία ότι πρέπει να περιοριστούμε βασικά στου 1,5 βαθμού. Ένα σημείο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς ε, εταίρους μας στην Προδευτική Συμμαχία. Έτσι λοιπόν ο μακροπρόθεσμος ε, στόχος ε, που έχουμε σημαίνει ότι αφού πολύ σύντομα φτάσουμε στο υψηλότερο βαθμό οι εκπομπές, μετά πρέπει πολύ γρήγορα να αρχίσουν να μειώνονται και να γίνεται και αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει το 2018 προκειμένου να καταφέρουμε να δούμε τι έχουμε πετύχει όσον αφορά τους δύο βαθμούς. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμεινε κάθε πέντε χρόνια να γίνεται αναθεώρηση. Και επίσης ζητήσαμε και διαφάνεια και λογοδοσία. Ξέρουμε ότι πρόκειται για τις βάσεις κάθε αξιόπιστης διεθνούς συμφωνίας, γιατί χωρίς συμφωνημένους κανόνες πολυμερός δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι οι χώρες θα φέρουν και τα αποτελέσματα για τα οποία δεσμεύτηκαν. Έτσι λοιπόν με τη συμφωνία αυτή οι χώρες νομικά δεσμεύονται να πετύχουν τι σημειώσει για τις οποίε έχουν δεσμευτεί. Αυτά τα στοιχεία αντιστοιχούν στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζουν και διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά τους στόχους που επιτυχάνουν οι χώρες. Τώρα, ε, όλα αυτά τα στοιχεία που θέλαμε περιλαμβάνονται στη συμφωνία, αλλά η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι ένα πακέτο αλληλεγγύης, όπως το λέμε, που περιλαμβάνει διατάξεις για χρηματοδότηση μέτρων υπέρ του κλίματος και αντιμετωπίζει τις ανάγκες λόγω των προσαρμογών, των απολειών, των ζημιών που γίνονται σε βάρος κάποιων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, και η Επιτροπή σας έχει αναγνωρίσει ότι το οικονομικό αυτό στοιχείο είναι στοιχείο κλειδί για τις διαπραγματεύσεις και πιστεύουμε και εμείς ότι θα πετύχουμε και είναι το 100 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο μέχρι το 2025. Όλες οι χώρες λοιπόν ενθαρρύνονται να προσφέρουν οικονομική στήριξη επιπλέον από τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει υπέρ των ε, αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών. Αξιόδημοι ευρωβουλευτές. Είναι μια ιστορική στιγμή και πρέπει να υποφεληθούμε από αυτή. Όμως μας περιμένει πολλή δουλειά. Αρχές 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί μαζί μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει προτάσεις για αποφάσεις από το Συμβούλιο μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενημερώνουμε πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο μέχρι το Μάρτιο του 2016 να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της COP21 προκειμένου κυρίως στα πλαίσια του κλίματος 2030 και του ενεργειακού πλαισίου να προετοιμαστούν τα επόμενα βήματα. Επιπλέον από την αξιολόγηση αυτή η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει και το νομοθετικό πρόγραμμα με εφαρμογή το, του πλαισίου για το κλίμα και για την ενέργεια του 2030. Τα επόμενα βήματα είναι να καλύψουμε και τους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Η Επιτροπή θα προτείνει λοιπόν μια προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε ένα μείον 40% στόχο. Αυτό θα συνδυαστεί βέβαια, θα και με τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την χρήση γης, την αλλαγή γης και την δασοκομεία, το λουλούκουφ όπως λέγεται. Οι σχεδιασμοί μας για τον επόμενο χρόνο όσον αφορά επίσης τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο στο έργο μας διότι θέλουμε η ενεργειακή αγορά να γίνει περισσότερο καθαρή και πιο αποτελεσματική. Η έρευνα και η καινοτομία επίσης είναι στο κέντρο της δράσης μας για το κλίμα με τον ορίζοντα 2020 που ήδη κάνει την διαφορά. Οι αλλαγές στο κλίμα και η εφαρμογή της COP21 σίγουρα θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο στο έργο μας αλλά και στις διεθνείς μας διαπραγματεύσεις και στο G20 και στο G7. Η κλιματική διπλωματία δεν θα σταματήσει θα λάβουμε υπόψη μα όλε τι πτυχές συμφωνία ε, του Παρισιού. Επίση, τα πλαίσια τη Σύμβαση για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών, και εκεί έχουμε δουλειά να κάνουμε. Το Παρίσι μα άφησε πολλά τεχνικά ζητήματα ανοιχτά. Μεταξύ άλλων, διατάξει όσον αφορά τη διαφάνεια και την ε, ε, λογοδοσία, τι στρατηγικές για το χαμηλό άνθρακα του 2050 και την συνέχεια από τη Λίμα στο Παρίσι όσον αφορά διάφορους μηχανισμούς ε, τεχνολογίας. Είναι αισθητική σημασία λοιπόν να συνεχίσουμε να οικοδομούμε και επιπλέον ικανότητες. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις προσπάθειες σας και για τη συνεχή σα συνεργασία. Καταφέραμε το Παρίσι να γίνει αυτό που θέλαμε υπέρ μιας παγκόσμιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και πιστεύω μπορούμε να ξεκινήσουμε πια με τον πρώτο γύρο των ομιλητών. κύριο Λίζε πρώτα, εκ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες και πιστεύω ότι δεν έχω καλύτερο τρόπο να συνοψίσω τους επένους προς τον κύριο Αρία Κανιέτε όσο ε, με τα λόγια του κυρίου Μπάς, του συναδέλφου, τα λόγια που χρησιμοποίησα την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι όταν όλοι οι βουλευτές συνενούν στους επένους ε, αποδεικνύεται ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Φυσικά ό,τι, λάμπει, δεν σημαίνει ότι είναι και χρυσός, αλλά η επιτυχία μας ε, στην COP21 είναι πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει βέβαια τις προσπάθειές της, αλλά έχει ένα μετάλλιο στο πέτο, ε, μια επιτυχία που έχει να επιδείξει στα χέρια της. Και πάνω σε αυτή μπορεί να χτίσει. Σε σχέση με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα σημαντικό βέβαια για την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στο Παρίσι, για τον χώρο των μεταφορών, ε, αέριων και θαλασσίων, μια και δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αυτές ε, στο, στη συμφωνία. Φαίνεται όμως το άρθρο 4, από ό,τι μου λένε, να υπάρχει μια έμεση έκκληση ή κλίση προς την ΙΚΑΟ και την ΙΜΑΟ ε, ίσως όμως ε, δεν έχω καταλάβει καλά. Θα ήθελα λοιπόν κάτι ευκρινήσεις από τον Επίτροπο και πάντως μετά τις επιτυχίες αυτές των Παρισίων μπορούμε να ασκήσουμε περισσότερες πιέσεις ώστε και η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειων Μεταφορών και η Διεθνής Οργάνωση ε, Θαλασσίων Μεταφορών να προχωρήσουν περισσότερο. Δεν μπορεί να δεσμεύονται όλα τα κράτη σε στόχους που βεβαίως εμείς θα θέλαμε να είναι και λίγο πιο φιλόδοξοι αλλά πάντως είναι πια εγγεγραμμένοι σε συμβατικά έγγραφα και οι, οι ε, υπηρεσίε αυτέ, το χώρο των εναέριων και των θαλασσίων μεταφορών, οι οργανώσει αυτέ, να μην έχουν φέρει κανένα καινούριο αποτέλεσμα. Ο κύριο Γκρότε. Ναι, βεβαίω ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία των Παρισίων και εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω, κύριε Επίτροπε. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πολύ καλή εκπροσώπηση, είχαμε και άλλε διασκέψει κόπο που είχαμε διαπιστώσει πω κάποια κράτη-μέλη προχωρούσαν να κάνουν δηλώσει ενώπιον των ε, ε, φακών της τηλεόρασης ε, μεμονωμένα. Δεν υπήρχε δηλαδή κλίμα ενωτικό. Ε, αυτή τη φορά βλέπουμε κάτι τελείω διαφορετικό και σα συγχαίρουμε. Ήταν πολύ καλέ οι επιδόσεις και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα διδάγματα τώρα από, το, από τη των Παρισίων είναι καταρχάς ότι με τη διπλωματία μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά. Και μάλιστα όταν είναι 195 τα συμβαλώμενα κράτη. Γι' αυτό και έχω την πρώτη μου ερώτηση λοιπόν σε σχέση με την ε, διπλωματία για το κλίμα που ξεκίνησε ο Λογόν Φαμπιούς ήδη από την αρχή αυτής της προσπάθειας, τι διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε και για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, ε, Δράσης, τι θα μπορούσαμε να διδαχθούμε ώστε να βελτιώσουμε την ε, κλιματική μας διπλωματία, πώς μπορούμε στη συνέχεια να αξιοποιήσουμε τις επιτυχίες αυτές. Δεύτερον, όσον αφορά τις ενέργειες και τις θαλάσσιες μεταφορές και τις συναντήσεις με την ΙΚΑΟ, βέβαια δεν ξέρω αν ε, δικαιούμαι να το πω γιατί ήταν και κλεισμένο των θυρών οι επαφές με την Κινέζικη Αντιπροσωπεία με άλλε είχαμε το δικαίωμα να μιλάμε πιο ανοιχτά, να βγάζουμε και φωτογραφίε κτλ. Με πάση περιπτώσει δεν θέλησαν ούτε οι Αμερικανοί να μα κακομάθουν ήταν σαν να βρισκόμαστε σε δύο διαφορετικούς πλανήτες λοιπόν σε σχέση με τις ανταλλαγές αυτές και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, μια και το έθιξε και ο Πέτερ Λίζε, τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα θέματα αυτά για να, για να ενισχύσει τις πιέσεις. Υπάρχει μια ε, χρονομέτρηση, starts the clock, υπαριθμών 1 που έχει ξεκινήσει. Τώρα έχουμε και την υπαριθμών 2 που αφορά τι ενέργειε και θαλάσσιε μεταφορέ. Τα κάνουμε λοιπόν για να πιέσουμε περισσότερο. Και πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αποστολή μια ομάδα στην ΙΜΑΟ. Γιατί παρεμποδίστηκε αυτό και υπήρξε μια αντιπαράθεση αρκετά έντονη που με ξενίζει. Ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει λοιπόν να δεχθούμε αυτή την ε, αδιαφάνεια σε επίπεδα ΙΜΑΟ και η καό, θαλασσιών και αερίων μεταφορών. Πρέπει να πιέσουμε για περισσότερη διαφάνεια, πρέπει να πιέσουμε για καλύτερους στόχους. Και βέβαια να είναι γνωστό τη σπάση τι κάνουν αυτές οι οργανώσεις. Η καό στο δεύτερο πυλώνα της ήταν μάλιστα εκείνη η οποία δήλωνε προθέσεις για περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος στο δεύτερο πυλώνα κλιματική αλλαγή, δεν είναι προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερε πιέσει. Κατά τα άλλα όμω και εν γέννη ευχαριστώ πολύ και πολλά συγχαρητήρια κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την πολύ καλή συνεργασία με την αντιπροσωπεία. Ήταν πολύ ευχάριστη κιόλα και ελπίζω ότι θα έχετε πολύ καλέ επιτυχίε και για το 2016, μια καλή χρονιά και καλά Χριστούγεννα φυσικά επί την ευκαιρία. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ, η κυρία Βυσνιέσκα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εάν κοιτάξουμε το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Ίσως ε, δούμε ότι είναι και κάπως αφιλεγόμενες οι επιτυχίες, γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις μεν σαν στόχοι για τους στόχους, αλλά δεν προβλέπονται συγκεκριμένε διαδικασίες για την επιτεύξη των στόχων αυτών. Και κάποιους στόχους τους ορίζουν τα ίδια τα μέρη βάσει της Συμφωνίας. Δεν είναι σαφές λοιπόν πώς μπορεί να ασκηθεί η πίεση προς τις συμβαλόμενες ε, πλευρές προς τα συμβαλόμενα μέρη για την επιτεύξη των στόχων. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ως προς την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. 55 χώρες ε, οι οποίες αντιστοιχούν μόνο στο 55% των όλων εκπομπών απαιτείται για να την κυρώσουν. Πράγμα το οποίο απαιτείται να την κυρώσουν για να τα θέσει λειτουργία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην συμπεριληφθούν σε αυτές ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα. Δεν ε, υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθυστερήσει και από πλευρά της την κύρωση και να περιμένει πρώτα οι Ηνωμένε Πολιτείε ή και η Κίνα να, την, ε, να κυρώσουν τη Συμφωνία των Παρισιών. Πράγμα το οποίο θα καθυστερούσε πολύ όλες τις εξελίξεις. Η δέσμευση άνθρακα επίσης από τους δρυμούς είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχετε κοιτάξει τη διάσταση αυτή, πώς μπορεί να ενισχυθεί δηλαδή ο ρόλος των δασών μας. Γιατί έτσι νομίζω μπορούμε να σβήνουμε περισσότερο και πιο γρήγορα τα επίπεδα των εκπομπών και να φτάνουμε ταχύτερα στους στόχους του περιορισμού των εκπομπών. Νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα δάση μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Ζουκέρμπαντι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω τον Πέτερ Λίσσα και τον Ματίας Γκρότε στα συγχαρητήρια. Προς εσάς κύριε Επίτροπε για τον ρόλο που διαδραματίσατε στο Παρίσι, κυρίως ε, το ρόλο του γεφυροποιού που διαδραματίσατε μεταξύ του πλούσιου τμήματος της Ιφιλίου με το λιγότερο πλούσιο, θα το πω έτσι. Και νομίζω ότι αυτό ε, σήμανε πολλά και για την επιτυχία μας στο Παρίσι. Μια και υπάρχει τώρα πια η συμφωνία λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, που ίσως είναι και πιο σημαντική ακόμη και αφορά την υλοποίηση. Πιστεύω ακράδαντα εν προκειμένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιολογήσει τις ε, συνέπειες της Συμφωνίας των Παρισιών ως προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια και για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εάν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχω συλλέξει, τον οδικό χάρτη για το χαμηλό άνθρακα του 2050 και αντίστοιχα του στόχους του 2030 για τις ε, κλιματικές αλλαγές αναφορίζεται το 80% αλλά αυτό δεν μπορεί να μας κατεβάσει κάτω από τους δύο βαθμούς αύξησης θερμοκρασίας ούτε καν, ούτε, και φυσικά ούτε κατά διάνοια να μας πάει στον 1,5. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ τι θεωρείτε ότι μπορεί να έχει σαν συνέπεια για την ευρωπαϊκή πολιτική το να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους του 1,5 βαθμού αύξησης για το 2050 και επίσης, μια και αναφέρθηκε νωρίτερα, η μέθοδος της ε, αναπενταετία αναθεώρησης Βέβαια προβλέπεται εδώ μια αναθεώρηση και των φιλοδοξιών για το 2018. Ε, τι σημαίνει αυτό για την Επιτροπή, πώς θα το χειριστεί το θέμα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε μια πρώτη αξιολόγηση το 2018 και να δει τι σημαίνει για τους στόχους μας για το 2020 και το 2030 αυτή η συμφωνία. Βέβαια αυτό ισχύει και για την διαρροή άνθρακα η οποία στηρίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα κάνει επαρκείς προσπάθειες ο υπόλοιπος κόσμος για τη συγκράτηση του άνθρακα. Τώρα μετά τη συμφωνία αυτό αλλάζει θεωρητικά. Άρα τι αλλαγές βλέπετε σε αυτό το θέμα. Και εν τέλει πρόεδρε, στο Παρίσι έγινε μια συμφωνία για τα 100 δις δολάρια ετησίως στη χρηματοδότηση για το κλίμα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα το δικό της μηχανισμό χρηματοδότησης που θα της επέτρεπε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο στόχο του των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Έχετε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένε, θα καταθέσετε ιδέες για έναν χρηματικό μηχανισμό ο οποίος αυτομάτως θα τροφοδοτεί το σχετικό ταμείο, τουλάχιστον δηλαδή το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριος Εκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Πέτροπε που είστε εδώ. Ξεκινώντας, ε, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή μετάβαση στο νέο έτος και πολλές επιτυχίες βέβαια στη δουλειά σας για το νέο έτος. Για την COP21 ε, και τις συμφωνίες της πρέπει να πω ότι έχω τις επιφυλάξεις μου για το εάν τα αποτελέσματα της COP21 είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας ε, πωλείται ότι είναι ή αν είναι δηλαδή μια μεγάλη ιστορική επιτυχία ή αν απλώς είναι μια ε, διευθέτηση. Γιατί και η πολιτική και ο τύπος χαιρέτησαν ε, την, τα αποτελέσματα της COP21 μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα αποτελεί μια καταγραφή της πραγματικότητας ε, και γι' αυτό έχω τις επιφυλάξεις μου εγώ μεγάλο κομμάτι των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα το παράγουν τομείς οι οποίοι δεν καταγράφηκαν στη συμφωνία, δηλαδή η μαζική γεωργική παραγωγή και η μαζική κτηνοτροφία. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν καλύπτονται και δεν υπάρχουν επαρκώς λεπτομερή μέτρα για τη συγκράτηση του διοξιδίου του άνθρακα στη συμφωνία η μέση αύξηση του πλανήτη θα πρέπει να περιοριστεί στο, σε ποσοστά λιγότερα, χαμηλότερα από τους δύο βαθμούς, αλλά οι στόχοι ορίζονται με τρόπο εθελοντικό. Και αυτό ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Δηλαδή οι κυρώσεις αποκλείστηκαν ήδη από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Και θα ήθελα κύριε Επίτροπε να μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δούμε στα επόμενα πέντε χρόνια ότι από χρόνο σε χρόνο συνεχίζεται η αύξηση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα αποδεδειγμένα. Εάν δούμε ότι στην επόμενη πενταετία αυξάνεται δυσανάλογα η κλιματική αλλαγή, δηλαδή εξελίξεις κλιματικές είναι προς τη δυσμενέστερη κατεύθυνση, πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ ξανά μαζί μας. Το έκανα ήδη στην Ολομέλεια και ο Πετρελίζε επίσης το επισήμενε. Ίσως σας έχουμε δώσει αρκετά συγχαρητήρια και ας περάσουμε τώρα στο τι περιμένετε από τους πρασίνους. Γιατί πρέπει να περιμένετε από τους πρασίνους γιατί αλλιώς μπορεί να εκνευριστείτε λίγο και δεν θέλω να σε εκνευρίσω πριν τα Χριστούγεννα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το πιο σημαντικό όταν συζητάμε κάτι τέτοιο είναι ότι κοιτώντα κανεί τι σημερινέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικό σα ισχυρισμό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται, πιστεύω ότι το σημαντικότερο το 2016 είναι να μπορέσετε να συνεχίσετε να κάνετε αυτόν τον ισχυρισμό, διότι αυτό ο ισχυρισμό ότι εμεί ηγούμεθα ε, γίνεται όλο και πιο ασαφής, ε, κυριότερα μετά από αυτές τις συμφωνίες του Παρισιού. Ε, αν θέλει λοιπόν η Ευρώπη να συνεχίσει να ηγείται και πιστεύω το θέλετε, θα πρέπει να δώσουμε και κάποια αποτελέσματα. Κοιτώντα τώρα τα σχέδια που έχουμε στο τραπέζι, δεν ε, παρέχουμε αρκετά ώστε να επιτύχουμε ε, τους δύο βαθμούς, ούτε καν τον, ένα, ούτε τον ενάμιση. Τώρα να λέμε να περιμένουμε μέχρι το 2018 μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα του IPCC. Αυτό δεν αρκεί γιατί ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που θα κάνουν την ανάλυση για το IPCC μπορούν να κάνουν την ανάλυση και για την Ευρώπη. Οπότε και εδώ θα μπορούσε να λάβει κάποια δράση η Ευρώπη. Κοιτώντα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και αυτοί θέλουν να ξέρουν τι σημαίνει αυτό πολύ κάτω από του δύο βαθμού ή ενάμιση βαθμό. Και εγώ πρέπει να σα πω ότι η βάση που χρησιμοποιούμε για όλε μα τι πολιτικέ δεν αρκεί. Διότι ο δικό χάρτη ε, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ε, με ορίζοντα το 2050 με μείον 20%, μιλάει για μείον 25% το 2020, δηλαδή ήδη πρέπει να κάνουμε περισσότερο για το 2020 και το μείον 40% μέχρι μείον 80%. Δεν είναι αρκετό για να πετύχουμε τους μείον 2, τους βαθμούς. Χρειαζόμαστε ένα νέο δικό χάρτη χαμηλών εκπομπών άνθρακα πέραν του 2020 ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η προσφορά βέβαια του μείον 30% και μου κάνει εντύπωση που δεν το αναφέρατε. Τι σημαίνει αυτό για το 2030 και τι σημαίνει για το 2050. Πρέπει να τα αναλύσουμε όλα αυτά ταχαίως πιστεύω. Και επίσης πρέπει να αλλάξουν κάποιες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα η μεταφορά που προτείνεται τώρα στο ETS από την τρίτη στην τετάρτη φάση αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τον σημερινό μας στόχο για το 2030. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να κάνει κάτι γι' αυτό και να πει αυτή η μεταφορά από το 30-40 πρέπει να ακυρωθεί. Το ε, Ταμείο Εξυγχρονισμού α, ουσιαστικά αποτελεί επιδοτήσεις για το ρηκτά καύσιμα μέχρι το 2030. Δεν νομίζω ότι αυτό δεν γραμμίζει τη με το Παρισί, δεν είναι. Οπότε ήθελα και σε αυτό το ταμείο να είμαστε λίγα πιο σκληροί από ό,τι υπήρξαν μέχρι στιγμή. Και όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα, πρέπει να αλλάξουμε του κανόνε ε, του εμπορίου. Γιατί πολλά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά λοιπόν που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε τι πολιτικέ μα. Και θα ήθελα μια πιο σαφή στάση από εσά ε, σχετικά σύντομα για το τι πιστεύετε για αυτέ τι αλλαγέ και τι θεωρείτε στην διαπραγματεύσει πιέζει, για παράδειγμα ω συνομοθέτε Πώ θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε πράγματι τι προτάσει σε σχέση με αυτέ που δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο. Ε, και κάτι τελευταίο, μια ερώτηση. Ε, πάντα κοιτώ με ευχαριστησή το λογαριασμό στο Twitter, αλλά ξέρετε τα tweets σα μερικέ φορέ δημιουργούν ερωτήματα. Την περασμένη εβδομάδα με μεγάλο ενθουσιασμό τουιτάρατε ότι για την ενεργειακή απόδοση θα προτείνετε πιο φιλόδοξου και πιο δεσμευτικού στόχου του χρόνου. Μπορείτε να είστε λίγο πιο ακριβεί. Τι σημαίνει αυτό. Και ελπίζω να μην πείτε το, τώρα θα πάμε στο μείον 30 αντί για μείον 27, γιατί εμείς ως κοινοβούλιο ε, θέλουμε να πάμε στο μείον 40. Ελπίζω να εννοείτε αυτό με το tweet σας. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα και ο Σπεντισίνη. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να πω πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ για τον λόγο. Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ κύριε Επίτροπε. Άκουσα πολύ προσεκτικά το όσα είπαν οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα λόγια σας και εσείς φυσικά έρχεστε να μας διηγηθείτε το όμορφο κομμάτι της συμφωνίας αυτής. Και μετά από τη διήγησή σας παρατήρησα ότι πολλές πολιτικές ομάδες, ειδικότερα οι μεγαλύτερες, κάπου χάρηκαν με τη διαπραγματευτική σας ικανότητα. Οπότε δεν θα σας αρεστήσει πιστεύω αν εγώ διαφωνήσω με αυτή τη χοροδία γιατί όταν φτάσατε εσείς εδώ και εγώ έφτασα εδώ συζητούσαμε πολύ για τη σύγκρουση συμφερόντων ε, με, επικεντρωθήκαμε σε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων ε, ενώ εγώ θεωρώ ότι από τη δική σας προηγούμενη εμπειρία στον κόσμο των επιχειρήσεων με την εμπλοκή σας στο τομέα του πετρελαίου θεωρώ ότι αυτή η σύγκρουση συμφερόντων που σας αφορά είναι πολιτική και τώρα αναδεικνύεται ε, η πραγματική σας θέση. Γιατί εγώ από τη δική μου πλευρά πίστευα ότι με την ευκαιρία αυτή δεν χρειαζόταν να εξετάσουμε τόσο το ζήτημα της ε, επιπλέον χρηματοδότησης των πολιτικών καταπολέμησης της ε, αλλαγής του κλίματος. Μιλάμε τώρα για ποσά ονομαστικά, αρκετά δισεκατομμύρια, αλλά στην πραγματικότητα είναι λιγότερα. Δεν ξέρουμε ποτέ αν θα φτάσουμε κάποιο τέτοιο αριθμό. Χρειάζονται ε, μεγαλύτερε μεγαλύτερες προσπάθειες αποφεύγοντας ε, τις πολιτικές που δημιουργούν την κλιματική αλλαγή. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε κάτι για τι επιχορηγήσεις ε, προ τα ορυκτά καύσιμα. Και αυτό δεν συνέβη. Στην Ευρώπη μιλάμε για 300, 300, 330 εκατομμύρια επιχορηγήσεις των ορυκτών καυσίμων ετησίως. Πολλά περισσότερα από ότι στην καλύτερο δυνατό σενάριο είχαμε προβλέψει για την πράσινη ενέργεια. Και αυτό είναι το θέμα και ε, σας ρωτώ, γιατί δεν κάνατε κάτι παραπάνω σε αυτό το τομέα. Πώς πιστεύετε ότι θα επιτύχετε πραγματικά ε, κάποιο καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή όταν έχουμε τέτοια αντίσταση από όσους έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στον τομέα του πετρελαίου και των ορειτών καυσίμων και συνεπώς δεν πρόκειται να αφήσουν ανοιχτό την εναλλακτική πορεία. Πώς πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με, την πρώτη, ε, ε, με τις πρώτες απαντήσεις. Οπότε δίνω αμέσω το λόγο στον κύριο Επίτροπο για την πρώτη σειρά απαντήσεων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μία δεύτερη σειρά ερωτήσεων. Αρκετούς που ζήτησαν το λόγο, ε, πολλοί συνάδελφοι. Οπότε και μετά από αυτέ τι απαντήσει θα έχουμε ένα τεράστιο πάλι γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και όλα μας τα μέλη που συμμετείχαν σε αυτό τον αρχικό ε, γύρο ερωτήσεων. Για να δούμε. Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ξέρετε, στο πλαίσιο των ΗΕ, η επίτευξη συμφωνιών είναι κάτι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο Δημιουργήσαμε τη σύμβαση του 1992 και χρειάστηκαν 23 χρόνια για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Διότι, ξέρετε, οι αποφάσει πρέπει να ληφθούν ομόφωνα. Έχετε 196 χώρε όλε μαζί. Και η ψηφοφορία τη του Βαλού έχει την ίδια αξία με την ψηφοφορία των ΗΠΑ. Αυτή είναι η δυσκολία σε αυτέ τι διαπραγματεύσει σε τέτοιε διαπραγματεύσει είναι σχεδόν αδύνατο να επιτύχει κανεί το 100% των στόχων. Αν με είχατε ρωτήσει την πρώτη ημέρα που ήμασταν στο Παρίσι, κατά, ε, κατά πόσο η συμφορία του Παρισιού θα ήταν αυτή που προέκυψε ότι ήταν, θα σα ε, έλεγα ότι φαίνεται αδύνατο δεδομένων των δυσκολιών. Σίγουρα. Υπάρχουν όμω πολλά στοιχεία. Ποιε ήταν οι προτεραιότητέ μα, ένα φιλόδοξο μακροχρόνιο ε, στόχο και ένα χρηματοδοτικό πακέτο. Αυτά τα πετύχαμε. Αλλά οι προτεραιότητες μας ήταν περισσότερες ακόμη. Κατά την άποψή μου έπρεπε να έχουμε συμπεριλάβει και τις εκπομπές από, την, από τις ενέργειες μεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Και το προσπαθώ μέχρι τελευταία στιγμή. Ξέρετε για την Ευρώπη οι θαλάσσιες και οι αεροπορικές μεταφορές ήταν ανέκαθεν παρούσες ε, στις ε, συνομιλίες μας με άλλους. Αλλά δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ε, ομοφωνία. Το ίδιο έγινε και με την επιχορήγηση των ορεικτών καυσίμων. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Είμαι υπέρ. Δεν έχει καμία λογική να δίνουμε επιχορηγήσεις και να τις διατηρούμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου είναι χαμηλή και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ε, απαλείψουμε σιγά σιγά τις επιχορηγίες προς τα ορεικτά καύσιμα και όσο το συντομότερο τόσο το καλύτερο αλλά αν ε, θέλατε να έχουμε μια τέτοια παράγραφο να πούμε ότι εξαλείφουμε τα ορεικτά καύσιμα μέχρι το 2020 αν είχαμε μια τέτοια παράγραφο 20 χρόνες χώρος μόνο θα συμφωνούσαν και χρειάζεται μια συμφωνία, είναι περίπλοκη Παρ' όλα αυτά στις συνομιλίες είδαμε το πνεύμα ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε πολιτικές καθαρής ενέργειας και να χρησιμοποιούμε χρήματα του προπολογισμού για να υποστηρίζουμε τα ρεκτά καύσιμα. Δεν έχει λογική. Το κίνημα της καθαρής ενέργειας βρίσκεται εδώ και θα παραμείνει. Οπότε θα χρειαστεί να περιμένουμε και η θέση της Κομισιόν είναι σαφής. Τα ρεκτά καύσιμα πρέπει να εξαλειφθούν. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφέροντος. Ε, είναι πολύ σαφής η άποψή μου για το τι πρέπει να, ποια πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Τώρα, ε, ποια διδάγματα μάθαμε στο Παρίσι. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να επιτυχούμε πλήρη ομοφωνία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη εμείς οι ίδιοι. Διότι εγώ μπόρεσα να βοηθήσω λίγο αλλά η Λουξεμβουριανή Προεδρία του, ε, του Συμβουλίου δεν ήταν πάντα εύκολο να επιτύχει ε, πλήρη ομοφωνία. Εμείς επιτύχαμε ομοφωνία στην εντολή διαπραγμάτευσης. Όταν ζητήσαμε ευελιξία διαπραγμάτευσης, το ζήτησα για το 1 ε, σημείο 5 από την Προεδρία, συμφωνήθηκε ομόφωνα. Εκεί εκφραστήκαμε με μία ενία φωνή. Το δεύτερο είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν μπορεί να έχει... Δεν μιλάω μόνο για το τμήμα για το κλίμα. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να εφαρμόσει σε ολόκληρο το έτος την ε, περιβαλλοντική ε, διπλωματία. Αυτό είναι για να ετοιμάσει την επόμενη κόπ και τις συνομιλίες στο Μόντρεαλ. πρέπει να έρθουμε σε επαφή και να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε πολλέ χώρε, κυρίω τι ε, λιγότερο αναπτυγμένε ε, χώρε. Με τι ΗΠΑ, ξέρετε, συναντιόμαστε καθημερινά με την Κίνα. Εντάξει, είναι διαφορετικό κόσμο, το παραδέχομαι, αλλά καθημερινά έχουμε επαφέ. Έχουμε τέτοιου είδου διάλογο. Αλλά με την Μπραζαβίλ, με το Κονγκό, με την Κάνα, με το Σουδάν, με την ε, Αιθιοπία δεν μιλάμε καθημερινά. Αλλά σε αυτέ τι διαπραγματεύσει ο λόγο όλων έχει σημασία και αυτό είναι από το σημαντικό δίδαγμα. Ότι και οι μικρέ χώρε είναι σημαντικέ και με αυτέ πρέπει να μιλήσει κανεί πρώτα και όχι μόλι δύο εβδομάδε πριν τι συναντήσει. Δεν μπορεί να επιτύχει κανεί συμφωνία μέσα στι τελευταίε δύο εβδομάδε. Οικοδομείται μια τέτοια συμφωνία. Οπότε πολλά είναι τα διδάγματα πρέπει να αποκομίσουμε. Όλοι σα ρωτήσατε την ίδια ερώτηση τι κάνουμε τώρα. Έχουμε τη συμφωνία στα χέρια μα, πού πάμε. Πρώτα απ' όλα να σα πω ότι έχουμε την πιο φιλόδοξη δέσμευση μπροστά μας ε, μετριασμού των εκπομπών. Αλλά δεν έχουμε την απαραίτητη νομοθεσία για να την πληρώσουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Οπότε αυτό το 40% τουλάχιστον που έχουμε στο τραπέζι είναι μακράν η πιο φιλόδοξη συμφωνία που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά ακόμα μας λείπει η νομοθεσία. Έχουμε το ETS, μιλάμε για μεταφορές, το κοινοβούλιο το γνωρίζει και η Κομισιόν πρέπει να χορηγήσει όλη την απαραίτητη νομοθεσία για να φτάσουμε αυτό το 40% γιατί δεν την έχουμε ακόμα. Τώρα πρέπει να περάσουμε από την οδηγία ανταλλαγής εκπομπών, το LULUCF. Κάποιος μίλησε για τα δάση για την τασοκομεία Ε, ναι, σίγουρα το ζήτημα της τασοκομείας μας αφορά ε, ε και, και διάφοροι άλλοι το ανέφεραν και κύριε Νιάσκα. Ε, ναι, ξέρετε το ζήτημα αυτό με τα δάση εντός του Λουλουσιέφ θα το συμπεριλάβουμε και στην οδηγία τη σχετική και θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο πηγαίνοντα πρώτα στην Πολωνία και μετά στη Φιλανδία και μετά στην Ιρλανδία γιατί αυτές είναι οι χώρες που έχουν προβλήματα με τα δάση και άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία με τις εκπομπές από εντατικές ε, ε, εντατική κτηνοτροφία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να συζητάμε χώρα προς χώρα για τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουν. Θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τα κράτη-μέλη για το επίπεδο προσπαθειών που πρέπει να, καταλάβουν, να καταβάλουν απλά για να επιτύχουν το 40%. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι το 40% είναι κάτι εύκολο. Δεν επιτυχάνεται τόσο εύκολο. Πρέπει να φτιάξουμε την νομοθεσία, να την θέσουμε σε ισχύ και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό ο φάκελο. Από την άλλη, το, Ευρωπο... το Συμβούλιο ζήτησε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Παρισιού και θα επανέλθουμε από αυτού το Μάρτιο. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να λάβει υπόψη το 1,5 τους 1,5 βαθμούς. Αυτή η μείωση του 40% του 2030 κινείται προς τους δύο βαθμούς εφόσον κάνει όλος ο κόσμος το ίδιο. Εμείς έχουμε και ένα παρελθόν και έχουμε και μια πορεία όπου μιλάμε για 80 με 90% μείωση των εκπομπών το 2050. Έχουμε λοιπόν ένα σαφή οδικό χάρτη για τους δύο βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε και το πώς θα λάβουμε υπόψη το φιλόδοξο στόχο του 1,5 ε, βαθμού ε, που υπάρχει στη συμφωνία, διότι υπάρχουν και οι ρήτρε αναθεώρησης ε, για καλύτερα αποτελέσματα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι αυτή η αξιολόγηση και μετά τη μελέτη αντικτύπου για τα εργαλεία που έχουμε, την οδηγία ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντα υπόψη τα διάφορα επίπεδα φιλοδοξιών. Δεν μπορώ να δεσμευτώ ούτε στο Twitter για καμία μεγαλύτερη φιλοδοξία πριν δω τη μελέτη αντικτύπου. Αυτό που είπα και το είπα στην ακρόασή μου, εδώ όταν ήρθα για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο, ότι η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε τουλάχιστον στο δεσμευτικό 30%. Το θυμάστε. Και δεν άλλαξα άποψη. με τους στόχους του 2030 και για το... Έχουμε ήδη πολιτικές ε, που έχουν τεθεί σε ισχύ τουλάχιστον μας το 2020 αλλά η Κομισιόν λαμβάνει πολύ ε, σοβαρά υπόψη την εκτίμηση δεκτή που θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, διαφανείς και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Οπότε θα αξιολογήσουμε τους εαυτούς μας και τη Συμφωνία του Παρισιού και επίσης θα κάνουμε τον πρώτο απολογισμό στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού ε, το 2018. Αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός. Και το να γίνει αυτός ο απολογισμός ε, δεν θα είναι συμφωνία, είναι απόφαση. Ε, γιατί η συμφωνία θα εφαρμοστεί από το 2021, οπότε έχουμε συμφωνήσει ότι θα κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό το 2018. Τότε λοιπόν το 2018 θα αξιολογήσουμε πώς εξέλιξαν τα πράγματα παγκοσμίω Έχουμε πολλές ευκαιρίες αυτή τη στιγμή. Το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει περισσότερες φιλοδοξίες από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Θα κάνουμε λοιπόν μια αξιολόγηση των πραγμάτων, θα κάνουμε την πρόταση που θεωρούμε εμείς καταλληλότερη και πιο ισορροπημένη και φιλόδοξη και μετά το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο. Και θα συζητήσει μαζί μας και εμείς με το Συμβούλιο. Ακούσαμε κάποια σχόλια για την θέση ισχύ της συμφωνίας και το πρόβλημα της νομικής δέσμευσης. Σύμφωνα με τη συμφωνία, όλα τα μέρη έχουν μια νομικώς δεσμευτική υποχρέωση να συμβάλλουν στο μετριασμό και να τον διατηρήσουν. Διαφέρει από το πρωτοκόλλο του Κιώτο. Ο στόχος μετριασμού ε, ε, επιβάλλει πρέπει να παραμείνει. Αυτό σημαίνει ότι όταν επικυρώσει κάποιο τη συμφωνία δεσμεύονται όλα τα μέρη να εφαρμόσουν εγχώρια ε, μέτρα μετριασμού ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Για τη μείωση των εκπομπών. Πρόκειται για μια δέσμευση να αναλάβει δράση κάθε μέρος ε, βάσει των στόχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτό αποτελεί μια στιβαρή βάση. Είναι σαφές ότι πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία. Έχουμε νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις και πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ταχεία συμμετοχή των ε, ΙΠΑ με, με πραγματική δράση. Είναι δύσκολο να περάσουν οι περιβαλλοντικοί νομοθεσίε στι Ηνωμένε Πολιτείε στο Γερουσία. Πρέπει να γίνει με εκτελεστική δράση και χρειαζόμαστε μια συμφωνία που να δεσμεύει τι Ηνωμένε Πολιτείε να διατηρήσουν του στόχου μετριασμού αλλά και να καταστήσει δυνατό για αυτούς να περάσουν από μια διαδικασία μέσω τη οποία θα μπορέσουν να ε, ε, εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά με αποτελέσματα. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Συζητούσαμε με τι ΗΠΑ για ένα έτο χωρί καμία κίνηση από πλευρά του και η ε, κίνηση τελικά ήρθε τι τελευταίε τέσσερι ημέρε τη τελευταία εβδομάδα. Ήταν εξαιρετικά περίπλοκο λοιπόν. Αλλά όπω είδατε με κάποια δουλειά επιτυχάνονται κάποια αποτελέσματα. Μια άλλη ερώτηση που ακούσαμε αφορούσε τη θέση σε ισχύ της ε, συμφωνίας και τα προβλήματα ε, της θέσης ισχύ συζητήθηκαν, πρέπει να σας πω, και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ορισμένε χώρες σε ορισμένες προτάσεις αρχικά έλεγε, αναφερόταν ότι η απόφαση θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μόνο σε ορισμένε χώρες ε, και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των εκπομπών. Τέλος, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για να είναι ουσιώδηση η συμφωνία θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό χωρών και ένας Συγκεκριμένο αριθμό εκπομπών. Οπότε λέγεται ότι θα τεθεί σε ισχύ ε, τουλάχιστον από 55 χώρε που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το 55% των συνολικών εκπομπών. Οι αριθμοί αυτοί επελέγησαν ώστε να διασφαλίσετε η συμμετοχή των μεγαλύτερων υπευθύνων εκπομπών. Ε, διότι η Κίνα, η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτές που πρέπει οπωσδήποτε να επικυρώσουν τη συμφωνία. 187 μέρη έχουν συμφέρει, 150 ηγέτες μίλησαν στη διάσκεψη, στην αρχή της δηλαδή. Όλα αυτά διασφαλίζουν ότι με τη συμφωνία αυτή θα μειωθούν ουσιαστικά οι εκπομπές. Οπότε ας ελπίσουμε ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα θα επικυρωθεί η συμφωνία αυτή. Τώρα, στην ε, Κοπεχάγη δεσμευτήκαμε με 200 εκατομμύρια για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναπτυγμένες συζητήσαμε κατά πώς θα επιτευχθεί το ποσό αυτό ή όχι. Αποφασίσαμε λοιπόν μετά στις Ηνωμένε Πολιτείες να υιοθετήσουμε μια μεθοδολογία όσον αφορά τις επιπτώσεις στο κλίμα για την προσαρμογή, για την μείωση για το μετρασμό οτιδήποτε τέλο πάντων έχει να κάνει με τι αλλαγέ όσον αφορά τι εκπομπέ και τι επιπτώσει στο κλίμα. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εξή. Είναι ότι τα περισσότερα ποσά δεν πηγαίνουν στην προσαρμογή. Πηγαίνουν στην μείωση, μετριασμό, mitigation. Θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο προς μια καλύτερη ισορροπία 50% μπορούμε να πούμε mitigation, 50% adaptation. Εύκολο είναι να το πει αυτό κανείς. Όμως η κύρια συζήτηση στο Παρίσι ήταν σαφής. Τα 200 εκατομμύρια θα είναι από την αρχή, από τις αναπτυγμένες χώρες. Μετά το 2020 οι αναπτυσσόμενες χώρες προχωράνε και αυτές στην τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει. Επιπλέον, όλες οι χώρες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν αναπτυσσόμενες χώρες, θα βοηθήσουν. Η Κίνα, η Σιγκαπούρη, Κορέα, που δεν ονομάζονται αναπτυγμένες, αλλά είναι οικονομίες αρκετά στεναρές. Θα βοηθήσουν και αυτές λοιπόν, τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα θα υπάρξουν πολλοί δωρετές. Το 2020 θα πρέπει να καθοριστούν ετήσιοι στόχοι. Πάντως δύο πράγματα είπαμε. Ότι θα αυξήσουμε το επίπεδο στήριξης. Ήδη δίναμε 56% πέρυσι. 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές και έχουμε δεσμευτεί να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Η Γερμανία, η Γαλλία, το Ενωμένο Βασίλειο έχουν δεσμευτεί για να ενισχυθεί αυτό το επίπεδο στήριξη στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο των ομιλητών. Καλό τους συναδέλφους να περιορίσουν τον χρόνο τους σε ένα με μισή λεπτά Ο Καρλ Χάιντς Φλόρενς πρώτος. Κύριε Επίτροπε, θα συμφωνήσω κι εγώ με χαρά στους επένους που εξέφρασαν οι συνάδελφοι προς το πρόσωπό σας. Ο Υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας βέβαια διαγραμμάτισε και εκείνος από πλευρά του ένα πάρα πολύ καλό και θετικό ρόλο. Το επισημαίνω. Ο Γιούντελ Μπέκε και ο κύριος Μέτλερ, οι δύο συνεργάτες σας επίσης, έχουν κάνει τεράστια δουλειά ιστορική σημασίας εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό είναι επιτυχημένη η διάσκεψη των Παρισιών, γιατί επιλέγει μια διαφορετική δομή, διότι άφησαν τα κράτη-μέλη τις εγωιστικές τους τοποθετήσεις και προχώρησαν σε μια γενικότερη λύση. Και αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία των Παρισίων. Τώρα στο παραπέντε σε σχέση με τα Χριστούγεννα μόλις πριν ε, τις διακοπές ε, και κυριολεκτικά στις 12 παρα 5 ε, δεν θέλω να κάνω επικριτικές τοποθετήσεις αλλά πρέπει να προσέξουμε πολύ κύριε Επίτροπε την κύρωση και πάνω απ' όλα υλοποίηση από τα αναπτυσσόμενα κράτη γιατί εκεί κινδυνεύουμε ιδιαίτερως ε, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά, εύχομαι κάθε επιτυχία, χρόνια πολλά καλά Χριστούγεννα και πολύ καλή υγεία. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σπαγνιού, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την ε, πολύ σημαντική δουλειά που κάνατε στο 15 μέρο αυτό προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η συμφωνία είσαστε ο ήρωας της COP21. Να, και ως απόδειξη εδώ έχουμε φοιτητέ από την Βόρεια Γαλλία που ήθελαν αυτή την τελευταία ημέρα εργασιών για το 2015 τον, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δουν τον Επίτροπο ο οποίος δεν πραγματεύτηκε αυτά τα θέματα με σάρκα και οστά. Και γι' αυτό και τους ε, δέχτηκα και τους έφερα στην συνεδρία σε μας σήμερα. Η συμφωνία λοιπόν αυτή που έχει, ε, μάλλον η συμφωνία την οποία έχει ζητήσει με τις ε, αποφάσεις του Κοινοβούλιο πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν ασφαλώς πολύ πιο φιλόδοξη. Βέβαια πολλές από τις προτάσεις μας περιλαμβάνονται στις ε, συμφωνίες των Παρισίων και είπατε κι εσείς ότι θέλετε να συνεχίσετε την προσπάθεια σε συνεργασία με μας το Κοινοβούλιο. Και εδώ νομίζω τρία σημεία θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε αυτήν την κοινή δουλειά. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν παρατηρητές και μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σε σχέση με τους προς επίτευξη στόχους και την ε, αναθεώρηση, αναθεώρηση του σχεδιασμού για το 2020, αναθεώρηση εφαρμογής για το 2025 και το καθεξής. Ε, άρα λοιπόν μέχρι την COP22 του Μαρακές δεν θα πρέπει αυτό το χρόνο που μας μένει να τον αξιοποιήσουμε και με βάση και τις εθνικές ε, συμβολές για να βελτιώσουμε την ε, συμβολή στον περιορισμό της παγκόσμιας δημοκρασίας. Επίσης τα 100 δις δολάρια και το ταμείο. Με τι μηχανισμό θα υλοποιηθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον, η αλλαγή οικονομικής ε, συμπεριφοράς. Ναι, έγινε λόγος για την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων κλπ. Βεβαίως και πρέπει να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα την ε, κυκλική οικονομία, να αποφύγουμε τη σπατάλη τροφή, μόνο να ενισχύσουμε την εφορορία στην γεω στην γεωργία και την κτηνοτροφία ε, και πολλά άλλα θέματα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιους στόχους για τα επόμενα χρόνια από πλευρά σας. Ευχαριστώ. Φαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και καλημέρα σας Επίτροπα. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνατε στην COP21 ε, και ευχαριστώ ιδιαίτερω για την υποστήριξη που προσφέρατε στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Όπω είπαν ήδη οι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, οι αέριες και θαλάσσιε μεταφορέ αποκλείστηκαν από την COP21 παρά τι πιέσει ε, που άσκησε και τόσο και το Κοινοβούλιο όσο και η δική σα Επιτροπή. Ξέρουμε ότι δεν, ε, δεν συνέπραξε, δεν ήταν συνεργατή βιώσιμη η ε, Διεθνής Οργάνωση Θαλασσίων Μεταφορών και μάλιστα προσπαθήσαμε να ρωτήσουμε και τον εκπρόσωπό της που ήταν παρόν στο Παρίσι, αλλά αποτελέσματα δεν ε, είδαμε. Ε, βρέθηκε βέβαια σε δύσκολη θέση. Πώς μπορούμε να μειώσουμε, κύριε Επιτροπέ, τις εκπομπές, τις θαλάσσιες μεταφορές, πώς μπορούμε να περιλάβουμε τον τομέα των θαλασσιών μεταφορών και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα UETS για, το, για τις εκπομπές και επίσης δεν μπορεί να επιβληθεί ένας φόρος για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα ανατόνο στους ευρωπαϊκούς λιμένες που θα χρηματοδοτούσε ένα ταμείο αποζημίωσης που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν στη συνέχεια οι ε, φορείς ε, που ασχολούνται με τις θελασσίες μεταφορές προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την αναπροσαρμογή τους ε, στις νέες συνθήκες ή φερειπή να υπήρχε μια δυνατότητα για επιλογή μεταξύ των δύο φυσικών συστημάτων. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Αφρόντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια σκέψη και δύο ερωτήσεις η σκέψη μου σε ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας η λέξη ανανεώσιμος εμφανίζεται μια φορά στις αιτιολογικές σκέψεις όταν μιλάμε για την ανάπτυξη της Αφρικής δεν υπάρχει λέξη άνθρακας, πετρέλαιο, ε, εξάλληψη του άνθρακα έχουν εξαφανιστεί όλες οι λέξεις αυτές έχουμε λοιπόν μια συμφωνία με διάφορους στόχους αλλά γραπτά δεν υπάρχει καμία καθαρή στρατηγική για την επίτευξη των στόχων. Και εσείς είπατε πολύ σαφώς και εγώ συμφωνώ, ότι επειδή ήταν 196 χώρες που κάθισαν γύρω από το τραπέζι, το αποτέλεσμα αυτό ήταν ήδη θετικό το ότι κάθισαν όλοι γύρω από το τραπέζι. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Αλλά σε τέτοιου είδου συμφωνίε αναγκαστικά πρέπει να επιτυγχάνεται κάποιο συμβιβασμό. Και είπατε εσεί ότι είναι αδύνατο να επιτύχουμε το 100% από μια τέτοιου είδου συμφωνία. Και ίσω γι' αυτό υποβαθμίστηκαν τόσο πολύ οι προσδοκίε και οι απαιτήσει από μια τέτοια συμφωνία που έπρεπε να είναι πιο ισχυρή, πιο αποφασιστική. Οι δύο μου ερωτήσει τώρα ε, μου κάνει έκπληξη ότι αντί για τη λέξη εξάλληψη του άνθρακα εμφανίζεται αυτός ο μηχανισμός αρνητικών εκπομπών, δηλαδή της δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα, που δεν γίνεται μόνο μέσω των δασών, μακάρι να ήταν έτσι, αλλά υπάρχουν και τεχνολογίες σε εξέλιξη που αφορούν τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και που δημιουργούν πολλές επιστημονικά. Ε, μεταξύ των επιστημόνων. Ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτές τις τεχνολογίες. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι τεχνολογίες θα λειτουργήσουν, ε, ότι εξελίσσονται όντως ε, υπάρχουν κίνδυνοι που δεν έχουμε αξιολογήσει πλήρως. Και η δεύτερη ερώτηση, πολλές φορές είπατε ότι είναι νομικώς δεσμευτική αυτή η συμφωνία. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς τι γίνεται αν μια χώρα υπογράψει αυτή τη συμφωνία και δεν την τηρήσει. Μπορείτε να μου απαντήσετε, να ξέρουμε τουλάχιστον τι σημαίνει πραγματικά το νομικά δεσμευτικό. Ναι, ευχαριστούμε ο κύριος Μπάλτσο. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Ναι. Έχω μια ερώτηση, Πρόεδρε. Ποιος είναι ο κύριος στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πήγε στην διάσκεψη των Παρισίων. Θέλαμε να δείξουμε πάλι ότι είμαστε πρωτοπόροι στην προστασία του κλίματος. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικός στόχος ή ότι επιτυγχάνεται γιατί είμαστε υπεύθυνοι του 9% των παγκόσμιων εκπομπών. Νομίζω ότι ο στόχος ήταν περισσότερο να υποδείξουμε τι είδους ε, στόχους μπορούμε να επιβάλλουμε στους άλλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, να δεσμευτούν σε συγκεκριμένους στόχους. Αυτό το καταφέραμε, γιατί τώρα βέβαια μπορεί να χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις, αλλά το 2016 θα εκλεγεί ασφαλώς ε, ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στις Ηνωμένε Πολιτείες και πρόεδρος ο οποίος δεν θα ακολουθήσει τις δεσμεύσεις του Ομπάμα. Τι θα γίνει λοιπόν στη συνέχεια. Επίσης τα 100 δις ε, δολαρίων που υποτίθεται ότι θα διαθέσουν οι ανεπτυγμένες χώρες, γιατί η Κίνα δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία αυτή. Θα τους δώσουμε χρήματα από αυτά τα 100 δις. Και η Ουγγαρία, για να το πω διαφορετικά, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρεθεί να χρηματοδοτεί την Κίνα, τη δεύτερη σε μέγεθος οικονομία, και μια χώρα με τεράστια αποθέματικά σε ε, συνάλλαγμα. Ευχαριστώ κύριο Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Και ασφαλώς θα βρείτε το χρόνο να ξεκουραστείτε μέσα στις διακοπές ύστερα από τις ξάγρυπνες εκείνες διαπραγματεύσεις. Θέλω να θυμίσω, μια και κάνατε και εσείς λόγο για την ακρόαση σας πριν από ένα χρόνο εδώ στο Κοινοβούλιο, για τους επικριτές σας, πόσο σκληρές ήταν οι τοποθετήσεις τους και πόσο βέβαια τώρα σας επενούν. Και, πα, και άξια νομίζω. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε πάνω απ' όλα να εξελιχθούμε σε ένα παγκόσμιο σύστημα περιορισμού των εκπομπών. Μπορεί η συμφωνία να έχει διατυπωθεί σε ένα κάπως συμβιλικό, με ένα συμβιλικό κάπως τρόπο, αλλά μπορούμε νομίζω και γι' αυτό σας ερωτώ εάν σκοπεύετε να αναλάβετε πρωτοβουλία για να δώσετε τον αρκτήριο λάκτισμα σε αυτή την ε, εξέλιξη, δηλαδή την ανάπτυξη ενός συστήματος ανταλλαγής ρήπων εκπομπών, αφού πια μπορούμε να πείσουμε τους εταίρους μας πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο φιλόδοξο σύστημα ανταλλαγής εκπομπών. Ο κύριος Πέτερλε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στο Παρίσι δεν πετύχαμε απλώς συμφωνία, πετύχαμε και περισσότερη Ευρώπη, οπότε κύριε Επίτροπε συγχαρητήρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως και για την προσωπική σας δέσμευση. Για την ελπίδα που μας δώσατε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Η εφαρμογή θα πετύχει μόνον εφόσον οι στόχοι είναι ελκυστικοί και αν ε, στηρίζονται με τις κατάλληλες στρατηγικές. Εγώ βλέπω δηλαδή εδώ μια μοναδική πραγματικά ευκαιρία, κυρίως αν καταφέρουμε με την Κίνα, την ε, Ιαπωνία και άλλες χώρες να ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή. Για την Ινδία, πιο συγκεκριμένα. Η Ινδία θα αναπτυχθεί οικονομικά όλο και περισσότερο. Δεν θα συνεισφέρει όμως την επίτευξη των στόχων χωρίς να έχει και μια στρατηγική, πράσινη στρατηγική, μια στρατηγική υπέρ της πράσινης οικονομίας. Πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βοηθήσουμε την Ινδία υπέρ μιας πράσινης οικονομίας. Με χαρά συμμετείχα στις συζητήσεις με την αντιπροσωπεία της Ινδίας στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι αυτά που λένε πάνε προς την ίδια κατεύθυνση που λέτε κι εσείς. Έπειτα, όσον αφορά τα ορυκτά. Η Ινδία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τον άνθρακα έτσι εν μία νυχτή. Το ζήτημα είναι ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να χρησιμοποιήσουν περισσότερο άνθρακα. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Ευχαριστούμε, ο κύριος Ντάνσκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε, τα αλλά Πράγματι είναι καλό να έχουμε περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερα παραδείγματα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πετύχει αποτελέσματα. Οπότε συγχαρητήρια και ευχαριστούμε για τα όσα πετύχατε την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ σύντομα τώρα. Αναφερθήκαμε στον εξωτερικό παράγοντα. Τι δηλαδή πρέπει να κάνουμε ώστε και άλλες χώρες στον κόσμο να εφαρμόσουν τα σχέδια τα οποία έχουν υποβάλει και να προχωρήσουν στην νομοθεσία τους. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σχέδια έχει ώστε η εσωτερική νομοθεσία των χωρών να αλλάξει έτσι ώστε να τίνουμε προς τον 1,5 βαθμό που έχει συμφωνηθεί. Τι θα γίνει λοιπόν και πώς θα μειωθούν τα αρνητικά αποτελέσματα με την νομοθεσία των χωρών μελών, γιατί αλλιώς υπονομεύεται ο στόχος και δεν θα πετύχει. σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δύο ερωτήσεις έχω για τη Γεωργιά. Πρώτον, σε τι βαθμό πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να έχουμε νέες πρακτικές, καινοτομία, νέες τεχνολογίες στη Γεωργία για τις καλλιέργειες ε, για περισσότερη ποικιλομορφία, στις καλλιέργειες για την ποιότητα του, της γης, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές από την καλλιέργεια και να προσαρμοστούμε επίσης στις κλιματικές αλλαγές. Πού βλέπετε εσείς τη μεγαλύτερη ευκαιρία όσον αφορά τη γεωργία. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει περισσότερε λεπτομέρειες όσον αφορά την ε, γεωργία από τις εθνικές είναι Ηνωμένε Πολιτείε και Ευστραλία. Αυτό σημαίνει ότι ή άλλες ε, αναπτυγμενε χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ και Αυστραλία. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει περισσότερο τι πολιτικές θέλει να ακολουθήσει. Ρωτάω λοιπόν, σε τι βαθμό και πότε μπορούμε να περιμένουμε νέες ρυθμίσεις για τη γεωργία προς αυτή την κατεύθυνση και επιπλέον Ποιος θα γίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Τίμερμανς ή ο κύριος Χόγκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Κίλωνεν. η κυρια κιλωνα Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέρφους. Κύριε Επίτροπε, θέλω να συνεχίσω για τις μεταφορές. Δεν με εκπλήσει που δεν υπάρχει ενθουσιασμός για τα όσα αποφασίζονται εκεί. Εσείς, κύριε Επίτροπε Κανιέτε, θα συνεχίσετε τις συζητήσεις με τον Επίτροπο Μπότς και στο Συμβούλιο με τις χώρες ε, μέλη για τις εκπομπές ώστε ο τομέας των μεταφορών να συμμετάσχει γι' αυτός περισσότερο στην όλη διαδικασία. Οι μεταφορές αποτελούν ένα πολύ βασικό παράγοντα επιβάρυνσης ε, της κατάστασης του κλίματος. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει να συμμετέχει και αυτός ο τομέας, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος... Ε, ο Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της γεωργίας και το ρόλο της, κύριε Επίτροπε. Δεν βλέπω αρκετές αναφορές στη γεωργία στη συμφωνία, γιατί βέβαια ξέρουμε ότι αυτή συμβάλλει ιδιαίτερα στην παραγωγή αερίων που επηρεάζουν τις κλιματικές αλλαγές. Και δεν ξέρω αν πρέπει να την βλέπουμε σαν μόνο επιβαρυντικό για τις κλιματικές αλλαγές παράγοντα ή και σαν ε, ευνοϊκό. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό να το εξετάσουμε και αυτό για να αποφεύγουμε επιβαρυντικές για τις κλιματικές αλλαγές εκπομπές αερίων από την γεωργία. Υπάρχει το θέμα της, των εκπομπών μεθανίου, φερειπίν από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες ή από την χρήση ε, αζωτούχων αερίων. Ε, αντίστοιχα όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και αν στις ΗΠΑ και στους άλλους μεγάλους παραγωγούς υπάρχει μια επιλογή για αϊφόρο γεωργία, κτηνοτροφία και τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες θα περιορίζουν την, ε, τις ε, συνέπειες για την κλιματική αλλαγή. Από την άλλη βέβαια θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις λύσεις εκείνες οι οποίες μπορεί να προωθήσουν την δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα με νέες πολιτικές και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να πιέσουμε, να μειώσουμε τις εκπομπές. Και δεύτερη ερώτηση, στα βιοκαύσιμα, όπου νομίζω ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε τα βιοκαύσιμα να παράγονται με το σωστό τρόπο. Γιατί αν παραχθούν με εισφαλμένο, ε, μπορεί να αντικαταστήσουν μεν ε, ως, ε, στην χρήση τα ορυκτά καύσιμα, αλλά μπορεί να κάνουν εξίσου μεγάλο κακό με αυτά. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Ευχαριστώ κυρία Εύη. Ναι, ευχαριστώ. Σύμφωνα απόλυτα με τα όσα ρώτησε ο συνάδελφος ο κ. και ελπίζω ο κ. Επίτροπος να μπορέσει να απαντήσει με ακρίβεια για όλα αυτά. Εγώ ήθελα να επικεντρωθώ στο ζήτημα του ETS, ε, της ανησυχία ότι χρησιμοποιώντας τέτοια ε, εργαλεία αγοράς για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ε, και χρησιμοποιώντας μοντέλα όπως το cap and trade, η ερώτησή μου είναι κατά πόσο αυτά είναι αποτελεσματικά. Έχουμε πολλές αμφιβολίες, ειδικότερα με το σενάριο των, της αγοράς ανταλλαγών εκπομπών διεθνώς που θα επέτρεπε την αγορά τίτλων εκπομπών με πιο ευνοϊκές συνθήκες ε, ώστε να ε, καταστήσει ε, αναποτελεσματικές τις επενδύσεις για μείωση των εκπομπών και καθιστώντας άχρηστο τα μέτρα για την αγορά που είχαμε σκεφτεί. Θα αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του ETS θα κάνετε κάποια ειλικρινή συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν αναλλακτικέ για αυτό το σύστημα ώστε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά το ζήτημα του διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γκαρδίνη. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα να συγχαρώ τον Επιτροπό για τις προσπάθειες που έχει καταλάβει, καταβάλει. Με ανησυχεί μια τάση που υπάρχει σε αυτή την Επιτροπή μονίμως, ε, ακόμη και οι πιο νέοι θέλουν να ξεκινάνε από το μηδέν τη συζήτηση. Σαν όλα αυτά τα χρόνια εμείς να μην κάναμε τίποτα εδώ πέρα, σαν να παίζαμε. Ε, σαν να παίζανε όσοι βρίσκονταν εδώ πριν από εμά και όσοι μας, θα μας ακολουθήσουν χωρίς ποτέ να λαμβάνουν σοβαρά τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει. Πιστεύω ότι αυτή η στάση είναι πεδαριώδης ε, και με ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί σε τελική ανάλυση και αυτοί εδώ βρίσκονται μαζί μας να δουλεύουν και κάθε φορά μας αναγκάζουν να πάμε πίσω και να ξεκινάμε από το μηδέν. Όπως αυτό το Σαββρό της Πενελόπης. Φτιάχνουμε κάτι με μεγάλες προσπάθειες, με πολλή κούραση, να συμφωνήσουν 28 χώρες, να συμφωνήσουν 196 στην ΚΟΠ. Ε, και ξαφνικά έρχονται αυτοί εδώ και δεν δείχνουν καμία απολύτως εμπιστοσύνη σε τίποτα και πρέπει να ξεκινάει κανείς από το μηδέν έτσι ε, θα μείνουμε πάντα σε ένα επίπεδο συζητήσεων, όπου ποτέ δεν θα προχωράμε ούτε κατά ένα βήμα. Ε, εγώ λοιπόν ήθελα να απευθύνω ένα αίτημα προς τον Επιτροπό ξανά να μας διατρεί ενήμερους για τις εξελίξεις των δεσμεύσεων των διαφόρων χωρών όπως τις παρουσιάζουν και μετά πώς προτίθεστε να ελέγχετε αποτελεσματικά την τήρηση των δεσμεύσεων. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι αν σταθούμε στην επιτυχία του Παρισιού, που ναι ήταν επιτυχία, και όπως ακούω εδώ στην αίθουσα πολλοί Ευρωπαίοι επιθυμούν να οθήσουν την Ευρώπη, ήδη κάνει πολλά, να αναλάβει ακόμα πιο αυστηρές δεσμεύσεις. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό, αν το κάνει μόνη της η Ευρώπη, αν έχει προχωρήσει υπερβολικά θα μείνει μόνη της Ξέρετε, ο ηγέτης βρίσκεται ένα, δύο, τρία βήματα μπροστά, όχι περισσότερα. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να συνεχίσει να είναι ηγέτηδα, αλλά να την ακολουθούν στενά από πίσω οι άλλες χώρες αλλιώς. Ε, ε, εμείς απλά θα καταστρέψουμε τη βιομηχανία αντί να σώσουμε το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Πόλουτσι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι σε τόσο δύσκολες εποχές για την Ευρώπη τα συμπερασμένα του Παρισιού έδειξαν ότι αν ενωθεί η Ευρώπη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον κόσμο. Μετά από πολλές αποτυχίες επιτέλους έγιναν σημαντικά βήματα προς τα εμπρός και μας αξίζουν συγχαρητήρια. Τώρα δεν πρέπει να ε, αποδυναμώσουμε τις προσπαθίες μας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Πώς θα προχωρήσουμε. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, ε, πάω στο σημείο από το οποίο ξεκίνησα στο Παρίσι. Παίξαμε πολύ καλά ομαδικά ε, ως Κομισιόν, ε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Αυτό το ομαδικό παιχνίδι και αυτή η σχέση και η επαφή μεταξύ, η στενή μεταξύ της, της Κομισιόν του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου πρέπει να αποτελεί κανόνα στο μέλλον. Δεύτερον, μετά το Παρίσι, για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσει που αναλήφθηκαν και για να μείνουμε φιλόδοξοι, δεν πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο να επιταχύνουμε τι νομοθετικέ διαδικασίε που εξαρτώνται από εμά, από εδώ, από το Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν. Και τρίτον, επί τη ουσία, πώ θεωρείτε ότι η Κομισιόν μπορεί να διευκολύνει όσον αφορά τι δεσμεύσει που αναλήφθηκαν ε, τα κράτη-μέλη, πώ μπορεί να διευκολύνει τα κράτη-μέλη λοιπόν για τι δεσμεύσει που ανέλαβαν. Ε, ευχαριστούμε, κύριο Σαρίνοβιτ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπο που βρίσκεστε εδώ. Ακόμη και αν ήθελα να σας συγχαρώ για τη συμφωνία, ε, παρότι θέλω να σε συγχαρώ για τη συμφωνία, συγγνώμη, έχω κάποιες δύσκολες ερωτήσεις. Σύμφωνα με τις εθνικές δηλώσεις προθέσεων, κινούμαστε προς τους 2,7 ή 3 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν είναι να πέσουμε στον 1,5 βαθμό, χρειάζεται, χρειάζονται ριζικές αλλαγές και επιπλέον προσπάθειες. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν προς εσάς είναι ποιος αναμένεται να το κάνει αυτό, αυτή την επιπλέον προσπάθεια. Ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κάνει τέτοια επιπλέον προσπάθεια αυτοβούλος. Ε, η δεύτερη ερώτηση που έχω αυτή η λίγη παραπάνω προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι για να αποδεσμευτούν επενδύσεις, να ενθαρρυνθούν οι επενδυτές για να επενδύσουν σε τεχνολογίες φιλικές προς το κλίμα. Το πρόβλημα όμως που με απασχολεί είναι ότι οι επενδυτές δεν είναι τυφλοί. Αντιλαμβάνονται ότι ενώ εμείς συζητάμε για 1,5 βαθμό, αυξάνουμε την κατανάλωση άνθρακα στη Γερμανία, ε, ανοίγουμε περιθώρια για το Nord Stream. Δεν μπορούν να συμφωνήσει η Γαλλία με την Ισπανία για την εξαγωγή της ε, ηλιακής ενέργειας κτλ. κτλ. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι τέτοιες ενδείξεις επηρεάζουν τη βούληση των επενδυτών να επενδύσουν σε τεχνολογίες φιλικές ε, προς το περιβάλλον ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5 βαθμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κ. Τζίσικε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και κύριε Καγκέτε. Συγχαρητήρια. Δεν ε, συνάδεται συμφωνία με 196 βαλόμενα μέρη κάθε μέρα. Πολύ μεγάλη επιτυχία σας. Πρέπει να έχουμε μια δεσμευτική βεβαίω συμφωνία που το λέμε είναι δεσμευτική αλλά έχει και τις αδυναμίες της και πρέπει να τις τονίσουμε. Δεν είναι συγκρίσιμες ε, οι ε, μειώσεις, ε, οι δεσμεύσεις για μειώσεις, πρέπει να υπάρχει συγκρισιμότητα, χρειάζεται διαφάνεια και για λόγους ανταγωνιστικότητας. Μιλούμε για την προστασία του κλίματος και για στόχους μειώσεως ε, της κλιματικής αλλαγής, αλλά υπάρχει και πίεση για το 2020 σε σχέση με την εγχώρια βιομηχανία. Γι' αυτό λοιπόν και με την Επιτροπή Βιανκόφσκα πρέπει να προσδιορίσετε συγκεκριμένα τι θα κάνετε στα επόμενα χρόνια. Η κυρία Σουίτσα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κανιέτσα και εγώ και να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που βλέπω επιτέλους ε, να λειτουργεί η διπλωματική, η περιβαλλοντική διπλωματία. Πρέπει βέβαια να δούμε τη συνέχεια, πώς θα τηθεί σε εφαρμογή η συμφωνία, αφού κυρωθεί από το 5% εκείνων που ε, συμμετέχουν κατά 50% στις ε, εκπομπές. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα όμως και ξέρω ότι τα έχουν διατυπώσει και άλλοι συνάδελφοι. Τι είδου κυρώσει θα επιβληθούν σε χώρες και επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Πρόκειται για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως όλους. Θα ήθελα να δώσω τα απαντήσει λοιπόν συγκεκριμένε πώς θα παρακολουθήσει την υλοποίηση της συμφωνίας η Επιτροπή. Κύριε Μακίνης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι κύριε Επίτροπε ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Ακούσατε για την γεωργία τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν εδώ στην Επιτροπή μας για τα βιολογικά ή την καινοτομία. Εσείς πού βλέπετε την ισορροπία όσον αφορά τη συνεισφορά της γεωργίας. Το θέμα της ασφάλειας τροφίμων που επίσης αναφέρεται στη συμφωνία μας ενδιαφέρει και θέλουμε να ξέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εσάς, τον Επίτροπο Χόγκεν και τους άλλους, τι συζήτηση γίνεται για τον προσανατολισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ήδη συμπεριλαμβάνεται μέτρα για το κλίμα στην ε, τελευταία μεταρρύθμιση, αλλά για το μέλλον τι προβλέπετε. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος λοιπόν. Και Έχετε ένα μεγάλο κατάλογο με ερωτήσει, οπότε σα ακούμε. Το πρόβλημα είναι ότι οι ερωτήσει. δεν είναι μάλλον ότι οι ερωτήσει είναι πολλές ή μεγάλε κτλ, αλλά ότι είναι δύσκολο να απαντηθούν. Είναι δύσκολε ερωτήσει. Τέλο πάντων, αρχίζω ευχαριστώντα σα για αυτέ. Η Γαλλική Προεδρία πρέπει να ξέρετε ότι έκανε εκπληκτική δουλειά όχι μόνο ο κύριος Φαμπιούς και οι συνεργάτες του, αλλά και οι συνεργάτες του κύριου Λαντ. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Ακούγαν τους πάντες, υπήρχε διαφάνεια στη διαδικασία. Και γι' αυτό και καταφέραμε να φτάσουμε σε τέτοια φιλόδοξα αποτελέσματα. Βέβαια, Προεδρία έκανε και κάτι που ξέχασα να πω και η Λουξεμβουριανή Προεδρία και η Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα έκαναν εξαίρετη δουλειά. Είχα συνεργαστεί στο παρελθόν με πάρα πολλές ομάδες. Ποτέ όμως δεν είχα συναντήσει συνεργάτες με τόσο ψηλές φιλοδοξίες και τόσο μεγάλη δέσμευση και αίσθημα καθήκοντος όπως οι συνεργάτες με τους οποίους δούλεψα για το COP21. Εξαιρετική βοήθεια μου προσέφεραν. Ε, τους ε, έλεγα κάτι και ερχόντουσαν με πολύ ξεκάθαρα αποτελέσματα, με ακόμα πιο φιλόδοξα από αυτά που είχα ε, θέσει εγώ. Δηλαδή πραγματικά τους ευχαριστώ. Ακόμα και οι ανακοινώσεις της Επιτροπής, γιατί συνήθως το χειρότερο που κάνουμε εμείς οι πολιτικοί, και βάζω και τον αυτό μου μέσα έτσι, τότε που ήμουν στη χώρα μου, είναι ότι δεν καταφέρνουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να περάσουμε το μήνυμα του τι κάνουμε. Οι πολίτες δεν καταλαβαίνανε τι κάνουμε. Λοιπόν, τώρα, το θέμα της επικύρωσης πρώτα. Η Επιτροπή δεν βιάζεται, φαντάζομαι οι χώρες μέρες έχουν διαφορετικά, διαφορετικές διαδικασίες. Αλλά βέβαια πρέπει όλα αυτά να γίνουν με διαφάνεια. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να επικυρώσουν, αλλά κύριο θα έρθει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε υπομονή. Η τροπολογία της Ντόχας το Κιώτο δεν έχει επικυρωθεί ακόμα από όλες τις χώρες μέλη. Πριν το Παρίσι δεν καταφέραμε να πετύχουμε την πλήρη επικύρωση του πρωτοκόλου του Κιώτο. Καταλάβατε. Υπάρχουν αργές διαδικασίες σε κάποιες χώρες, υπάρχουν πολιτικά προβλήματα σε άλλες. Ε, πάντων, ελπίζω ότι τουλάχιστον το Κιώτο θα επικυρωθεί. Γι' αυτό βιάζομαι. Για το άλλο έχουμε καιρό να συζητήσουμε για τις ημερομηνίες κύρωσης. Τώρα ο κύριος ε, Πανιό. Στις συμφωνίες και για τους ανθρώπους οι οποίοι θα αποφεληθούν και για τους φοιτητές που φέρατε. Εμείς προσπαθούμε να παρουσιάσουμε όσο γίνεται καλύτερα τον κόσμο τη συμφωνία. Εδώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Αλλά είναι δύσκολο να εξηγηθεί πλήρως. Στηρίζω πάντως τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αυτές είναι πολύ σημαντικές. Πάντως μια τέτοια συνεργασία λειτουργεί καλά. Για τις αναθεωρήσεις τώρα. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλές διαδικασίες απολογισμού αξιολόγηση. Όταν αξιολογούμε τις επιπτώσει τη συμφωνία cop COP21, αυτό σε πρώτο στάδιο θα γίνει στο Ερεινό Συμβούλιο. Τότε θα δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει παγκοσμίω και θα δούμε τι μπορούμε να προσαρμόσουμε. Πάντω, η πιο βασική ημερομηνία είναι το 2018. Τότε θα γίνει παγκοσμίω αυτή η αξιολόγηση. Τότε θα δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε στο μέλλον. Το 2018 θα καταλάβουμε συνολικά την κατάσταση. Αν μείνουμε στο 3,8 στο 4,7 θα είναι business as usual. Αν όμως δούμε ότι έχει αλλάξει και δεν είναι ο μέσος όρος αυτός 3,8 με 4,7 αλλά είναι 3 η αύξηση δηλαδή της θερμοκρασίας, εντάξει θα είμαστε πάνω από 2 βέβαια. Αλλά το 2018 όλοι θα πρέπει να δούνε πώς θα ανεβάσουμε τις φιλοδοξίες μας. Προηγουμένως πρέπει να εκτιμήσουμε την εφαρμογή των πολιτικών μας, πόσες χώρες όντως εφαρμόζουν τους συμβιβασμούς και τους στόχους, πρώτα εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις νύχες στον υπόλοιπο κόσμο. Ο κύριος Περνιό με ρώτησε για τη χρηματοδότηση. Τα 100 δισεκατομμύρια φυσικά και πρέπει να τα δώσουμε τα 100 δισεκατομμύρια είναι επιπλέον από την στήριξη όλων των χωρών μελών. Γιατί έτσι κι αλλιώ τέτοια πολιτική χρηματοδότηση μέτρων υπέρ του κλίματο έχουν σε εθνικό επίπεδο όλε οι χώρε μέλη. Αυτά τα χρήματα είναι επιπλέον από αυτά. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε με δημόσιο χρήμα την ε, προσαρμογή και την μείωση των εκπομπών γενικά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εξυπηρετούμε τη Συμφωνία του Παρισιού και να στηρίζουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Το Ταμείο Προσαρμογής φτιάχτηκε από το Κιώτο, άρα έχουμε πολλά οικονομικά μέσα. Αλλά πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Και εμείς από την Επιτροπή, αλλά και οι χώρες μέλη. Εδώ μπορούμε να πετύχουμε βελτιώσεις, κυρίως γιατί στη διαδικασία αξιολόγησης και απολογισμού δεν ε, αντιμετωπίζουμε μόνο το θέμα για την προσαρμογή, για τον μετριασμό, τη μείωση, δηλαδή adaptation and mitigation, αλλά ε, η αξιολόγηση θα γίνει και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μέτρων. Θα δούμε τι έχει εφαρμοστεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέχρι τότε, στην κάθε δηλαδή αξιολόγηση που θα κάνουμε. Τώρα, πολύ αναφέρθηκαν στις μεταφορές. Εδώ είναι σαφές ότι η Γεωργία και οι μεταφορές που δεν καλύπτονται πλήρως από την ε, συμφωνία εξαιτία της ιδιαίτερης φύσης τους, άλλες χώρες είναι υπέρ των αναλλακτικών πηγών ενέργειας, ε, για... έχουν άλλες πολιτικές στις μεταφορές σε άλλη βάση πολυμερή πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Σήμερα μιλάμε για πέντε. Αν να μειώσουμε τις εκπομπές σε όλους τους τομές, τομείς, το 2000 50, η αεροπορία για παράδειγμα μεταφορές θα είναι υπεύθυνη για το 33%. Άρα είναι εκπομπές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ρητή μνήα, το ότι χρειάζεται δράση είναι προφανές και είναι κάτι που πάει πιο μακριά από το Παρίσι. Υπάρχει ένας διεθνής ε, στόχος, υπάρχει το 1,5, 1,5 βαθμοί και όλοι οι τομείς πρέπει να συνεισφέρουν με ένα δίκαιο τρόπο. Το 2016 θα είναι έτος κλειδί για τους τομείς αυτούς. Και στην ΙΚΑΟ πρέπει να παρέμβουμε. Σήμερα κάποιος με ρώτησε για τη συνεργασία μου με τον Επίτροπο Μπέρκ. Πριν έρθω, μιλήσαμε για να συνδυάσουμε τις μεταφορές με το κλίμα στο Νικάο ακριβώς. Άρα, διπλωματικά πρέπει να δραστηριοποιηθούμε με χώρες της Αφρικής, Σαουδική, Αραβία κλπ και πρέπει να χτίσουμε συμμαχίες πριν πάμε στο Μόντρεαλ. Το σύστημα διακυβέρνησης είναι πολύ ιδιαίτερο και ένα από τα πράγματα τα, οποία συζήτησα με την κυρία Μπόρκ είναι πώς θα συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το θέμα αυτών των εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό. δεν κάνουμε τίποτα, το 2050 θα έχει αυξηθεί πάνω από 30% το ποσοστό του τομέα στις εκπομπές. Άρα πρέπει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και να συνεχίσουμε με τις καλές πρακτικές που έχουμε χτίσει μέχρι τώρα. Επίσης, είχαμε και κάποιους οι οποίοι με ρώτησαν για τις στρατηγικές που πρέπει να αναπτύξουμε. Έχουμε συμφωνία για το που χρειαζόμαστε στρατηγικές. Κοιτάξτε, έχουμε τη συμφωνία και έχουμε και όλους τους ε, δείκτες που παρουσιάζουν οι χώρες μέλη. 40% βασίζονται στις ανανεώσιμες. 30% λίγο πολύ επίσης. Δηλαδή η κάθε χώρα μπορεί να έχει διαφορετικό καθεστώς, ξεκινάει από αλλού και υπάρχει και θέμα Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε πρώτον ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσουμε τις φιλοδοξίες μας. Θέλουμε νέους στόχους. Υπάρχουν τρίτες χώρες, αν διαπιστώσουμε ότι δεν τηρούν τους στόχους, ότι δεν εφαρμόσουν την νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα η Επιτροπή θα πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο, εφόσον δεν υπάρχει δράση από τις χώρες μέλη. Τώρα για τρίτες χώρες. Κοίταξε, πρώτα εμεί λοιπόν πρέπει να βάλουμε τάξη στα δικά μας πριν πάμε στο διεθνέ επίπεδο. Γιατί στο Κιώτο υπήρξαν ε, παραβιάσεις. Οι 28 από 38 χώρες ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, στο Κιώτο. Εδώ όμως η διαφάνεια, η συμμόρφωση και η εφαρμογή είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα εδώ δεν είναι τόσο να μιλάμε για ακυρώσεις, όσο να μιλάμε για την αξιολόγηση, οπότε θα βλέπουμε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν μείνει πίσω για να τις βοηθήσουμε και θεσμικά και αλλιώς να προχωρήσουν, είτε πρόκειται για την πραγματογνωμοσύνη που θα προσφέρουμε, να βοηθήσουμε για την εφαρμογή ίσως με ε, κάποιες ομάδες ε, που θα φτιάξουμε ώστε να προχωρήσουν να επικεντρωθούν στα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουν και έτσι να καλύψουν την καθυστέρηση και τη διαφορά. Πάντως το Παρίσι είναι μια επίσης πολιτική διαδικασία. Αν δεν πετύχουμε θα υπάρξουν και πολιτικές συνέπειες σε εθνικό επίπεδο. Κάτι που δεν πρέπει να υποτιμάμε. Όταν αρχίσει η δράση θα υπάρξουν χώρες οι οποίες θα τα καταφέρουν και άλλες που δεν θα τα καταφέρουν. Όμως η κοινή γνώμη θα πιέσει. Όλος ο κόσμος θέλει καθαρό αέρα, καθαρή ενέργεια. Δείτε στην Κίνα. Η Κίνα πριν το 2030 θα φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και μετά θα αρχίσει η μείωση. Άλλες χώρες πολύ πιο γρήγορα. Γιατί, και η Κίνα ίσως, γιατί, γιατί σε εθνικό επίπεδο τη συμφέρει. Άρα δεν πρόκειται μόνο για την νομική υποχρέωση που αναλαμβάνουν οι χώρες μέλη, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να προχωρήσουν με τις φιλοδοξίες μας και στο Κιώτο. Εμείς ήμασταν φιλόδοξοι, όχι όμως ο υπόλοιπο κόσμος. Τώρα υπάρχουν τα ίδια επίπεδα φιλοδοξίας από όλου. Υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με τη βιομηχανία. για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ένα από τα καλά, τα θετικά που είδαμε, είναι ότι υπάρχει μια θετική τάση για την αγορά αυτή, για, την, για το εμπόριο αυτό εκπομπών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε σε ένα μεγάλο βαθμό πάνε προς την ίδια κατεύθυνση και η Κορέα. Και άλλες χώρες σκέφτονται αυτό το σύστημα εμπορίας εκπομπών για να έχουμε μια παγκόσμια αγορά άνθρακα. Οι αγορές θα συνδεθούν πολύ γρήγορα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ο καλός τρόπος να προχωρήσουμε. Με διαφορετικούς μηχανισμούς, αναφέρθηκε και ο φόρος για τον άνθρακα μόλα, τα προβλήματα που δημιουργούνται γίνονται υπολογισμοί για το πόσο μπορεί να συμπεριληφθεί η ευθύνη για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε κάθε προϊόν. Οι αγορές άνθρακα. Κάναμε σφάλματα στο παρελθόν. Τα διορθώσαμε. Το Κοινοβούλιο τώρα έχει την ευθύνη για να προχωρήσει περισσότερο. Διότι αν έχουμε μια παγκόσμια αγορά άνθρακα, τότε θα υπάρχουν ισότιμες συνθήκες για όλους. Πρέπει βέβαια να είναι συμβατή η στόχη μας με τον βιομηχανικό στόχο του 20%. Η συνεργασία πάντως με την Επίτροπο Μπέρκ ήταν εξαίρετη, όπως και με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανένα πρόβλημα. Το σώμα των Επιτρόπων το τωρινό έχει πολλές αρμοδιότητες, ο κύριος Σέσκοβιτ συντονίσει τις ομάδες, συνεργαζόμαστε και κάνουμε καλή δουλειά πραγματικά. Στα πλαίσια αυτά. Λοιπόν, με ρωτήσατε και για τη Γεωργία. Όπως καταλαβαίνετε, με τον Επίτροπο Χόγκαν συνεργάζομαι πολύ. Γιατί πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με το Λούκουφ, πώς θα προχωρήσουμε με την Γεωργία γενικότερα και αυτά τα συζητάμε μεταξύ μας οι δυο μας πριν πάμε στο σώμα των Επιτρόπων. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την γεωργία, της ε, λεκάνες αποθήκευσης, πώς ε, θα προχωρήσουμε με την δασοκομεία, τι γίνεται με την καινοτομία, πώς μπορούμε να στηρίξουμε με τον ορίζοντα 2020. Είμαι στην Ταϊλάνδη, στη Νέα Ζηλανδία, υπάρχει πολλή καινοτομία για να μειώσουμε τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα στις χώρες αυτές. Στο μέλλον, για τη νέα κοινή γεωργική πολιτική, φυσικά και θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ε, την δράση υπέρ του κλίματος. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συμφιλιώσουμε την ασφάλεια τροφίμων, πώς θα ταΐσουμε τον κόσμο δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο βέβαια εξάγουμε και πώς θα τα συνδυώσουμε αυτό με τη δράση μας υπέρ του κλίματος. Το μέλλον η κοινή γεωργική πολιτική θα απαιτεί τη συζήτηση για δράσεις για το κλίμα. Τι άλλο. Τι γίνεται με την εθνική νομοθεσία, με τις εθνικές συνεισφορές, τις δεσμεύσεις δηλαδή για την συνεισφορά της κάθε χώρας. η ενεργειακή απόδοση είναι το μέσο στον οποίο αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα προβλήματα. Υπήρξαν ερωτήσεις επίσης. Α, Ινδία. Ινδία. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ινδία. Ινδία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα οικονομικά, σίγουρα. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν αλλά θέλουν να αναπτύξουν και μέτρα για ανανεώσιμε πηγές ενέργεια. Έχουν μεγάλη φιλοδοξία και ζητούν τη στήριξή μα ε, όσον αφορά την τεχνολογία αυτή. Όπως προχωράνε με τον ε, άνθρακα, θέλουν να αποσύρουν παλιές βιομηχανικές μονάδες, αλλά εμείς αυτό που στηρίζουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τις ε, λεκάνες αποθήκευσης άνθρακα, την αποθήκευση άνθρακα, γιατί έχουμε την τεχνολογία για να απομονώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα και να το αποθηκεύσουμε σε λεκάνες. Το θέμα είναι οικονομικά πώς θα ε, μπορούμε να το κάνουμε πράγματι και τα ποσοστά. Πάντως μπορούμε να πετύχουμε τον ανάμιση βαθμό μόνο αύξηση της θερμοκρασίας κατά μέσο όρο εφόσον προχωρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν την τεχνολογία αυτή και να συνεργαστούμε με τις χώρες Καναδά, Αυστραλία, Κίνα που στηρίζουν αυτή την τεχνολογία και να έχουμε στο τεχνολογικό τομέα συνεργασία μαζί τους. Απ' την άλλη πλευρά, τι γίνεται με την εθνική συνεισφορά και τα μηνύματα που μας φτάνουν για τις επενδύσεις. Αν διαβάσετε τις εκθέσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας για την Ενέργεια, ναι, όντως δεν φτάνουν οι συνεισφορές αυτές για τους δύο βαθμούς. Πρέπει να γίνει μεγάλη αλλαγή και η κυκλική οικονομία σίγουρα θα βοηθήσει πολύ στις πρακτικές διαχείρισης. Οι επενδύσεις χρειάζονται για από τις 187 χώρες είναι 3 5 δισεκατομμύρια για τις ανανεώσιμες. Υπάρχουν τα μηνύματα από τα Ηνωμένα Έθνη. 187 χώρες που λένε αυτό θα κάνουμε για το ενεργειακό μείγμα. Τεράστια ευκαιρία αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό και εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τις οδηγίες μας και για τις ανανεώσιμες και για την ενεργειακή απόδοση, ώστε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο επίπεδο που θέλουμε. Αυτές ήταν... Α, άλλη μια ερώτηση για τη Γεωργία. Για τα βιοκαύσιμα ήμουν υπεύθυνο κάποια εποχή. Σίγουρα πρέπει να στηρίξουμε την οικολογική παραγωγή. Ήμουν υπουργό τότε και είχαμε φτάσει πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια. Το πιο σημαντικό είναι όμως να καταλαβαίνει ο καταναλωτής διαφορά. Υπάρχουν χώρες που εκτιμάται πάρα πολύ ο οικολογικός παράγοντας και τα βιολογικά. Αλλού όχι. Σε άλλες χώρες όχι. Για τα βιοκαύσιμα κάναμε σφάλματα στο παρελθόν που δεν πρέπει να επαναλάβουμε στο μέλλον. Αλλά υπάρχει μεγάλη ευκαιρία εδώ για τα βιοκαύσιμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εισαγάγει την κατάλληλη νομοθεσία με την γνωστή διαδικασία για να μην κάνουμε τα ίδια σφάλματα. Δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα προσπαθώντας να λύσουμε κάποιο άλλο. Ε, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Κάποιος αναφέρθηκε στους μηχανισμούς της αγοράς και τα προβλήματα που έχουμε το σύστημα εμπορίας του του άνθρακα. Στο Παρίσι προσπαθήσαμε να πετύχουμε συμφωνία έτσι ώστε οι μηχανισμοί της αγοράς να περιλαμβάνουν καθαρή ενέργεια και προσπαθήσαμε τους μηχανισμούς αυτούς να τους χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε και το περιβάλλον και το κλίμα και να μην παραμείνουν κενό γράμμα. Θα προσπαθήσουμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο. Στις επόμενες διασκέψεις COP θα φροντίσουμε να υπάρξει κάτι θετικό ώστε να υποφεληθούν όλοι να είναι υπέρ του περιβάλλοντος. Κάποιος ρώτησε τι θα γίνει με το σύστημα εμπορίας διοξιδίου του άνθρακα. Θα ενημερώσουμε την Επιτροπή σας για το πώς έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα το σύστημα αυτό ETS και πώς θα προχωρήσει. Θα σας δώσω αυτά τα στοιχεία. Κύριε Γκαρδίνη, εσείς εξηγήσατε πώς θα ελέγξουμε τη συμφωνία και τους συμβασμούς. Η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αξιολόγηση που θα γίνεται κάθε τόσο. Ακόμα και δεν υπάρχει το naming and shaming, παρόλα αυτά δημιουργείται πίεση από την κοινή γνώμη η κλιματική δράση ανανεώσιμες πηγές είναι κάτι που στηρίζει κοινή γνώμη. Και δεν είναι δυνατόν να το γνωρίσουν αυτό οι πολιτικοί, γιατί τότε η κοινή γνώμη θα τους τιμωρήσει. Σε ελάχιστε χώρες δεν υπάρχει ισχυρή θέση από την κοινή γνώμη. Ή τέλος πάντων να μην πω από την κοινή γνώμη, από τη, τους εθνικούς πολιτικούς, τις ΗΠΑ για παράδειγμα. Με το σύστημα όμως που έχουμε εφαρμόσει η αξιολόγηση αυτή, αυτό το peer review, τα στοιχεία δηλαδή ώστε να αυξηθούν οι φιλοδοξίες υπάρχει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Οι διάφοροι εταίροι πολλές φορές πάνε πιο γρήγορα και πιο μακριά από τη ίδια πολιτική. Για παράδειγμα για την καθαρή ενέργεια είναι πραγματικότητα και γίνονται επενδύσει όλο και περισσότερε και θα γίνονται και οι θέσεις απασχόληση που εξαρτώνται από τέτοιου είδου ε, πολιτική είναι επίση κάτι πολύ σημαντικό για όλου και αυξάνονται. Πάμε πιο γρήγορα πιστεύω στην πραγματικότητα από ό,τι πάνε οι εθνικέ δεσμεύσει για εθνική συνεισφορά. Συνεργασία, τι άλλο. Α, ναι. Ο κύριος Τσέροβιτς με ρώτησε κάτι. Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε τίποτα, θα είμαστε στο 3,7 με 4 και αύξηση στη θερμοκρασία. Οπότε αυτό που πετύχαμε στο Παρίσι, εφόσον βέβαια εφαρμοστεί πλήρω, θα βοηθήσει πολύ. Και τώρα πρέπει να δούμε πώς από το 2 θα αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας στον 1,5 μόνο βαθμό να δούμε πρώτα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να τίνουμε στον 1,5 βαθμό αντί για το 2 και μετά θα δούμε τι μπορεί να κάνει ο υπόλοιπο κόσμο για τι. κυρώσει σα. Είπα. Τώρα αν ξέχασα κάτι ζητώ συγγνώμη έτσι. Πείτε μου τι ξέχασα και ευχαρίστω να σα απαντήσω. Αλλά τα στοιχεία, όπω είπα, θα σα τα δώσω για το σύστημα εμπορία διοξιδίου του άνθρακα. Τι γίνεται και με τι επενδύσει εκεί κλπ. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις σας. Happy for the result of the uh, climate meeting in Paris and uh... και συγχαρητήρια και πάλι για το Παρίσι. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας με την επόμενη 14 Ιανουαρίου. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά.